Buonasera a tutti. Καλησπέρα σας. Saluto le interpreti. Χαιρετίζει τους διερμηνείς ο Πρόεδρος. Buonasera a tutti, innanzitutto voglio Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του Bundestag, τον κύριο Μάικλ Γκόλτμαν, καθώς και ολόκληρη την αντιπροσωπεία του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Iniziamo con qualche piccola variazione dell'ordine del giorno αρχίσουμε με κάποια μικρή αλλαγή της ημερήσιας διάταξης λόγω των ωραρίων πτήσεων των ειδικών, των εμπειρογνωμών που θα παρουσιάσουν την μελέτη για την απελευθέρωση του δικαιώματος εγκατάστασης. Ε, θα πρέπει να αλλάξουμε κάπως την ημερήσια μας διάταξη. Αύριο θα μιλήσουμε για την έκθεση του Αντιπροέδρου Βιζεβόσκη και μετά θα αναβάλουμε την ε, μελέτη, την παρουσίαση της μελέτης αυτής. Κατά τα λοιπά μένει, στην, μένει ίδια, εκτός από την παρουσίαση του Λουίς Καπούλα Σάντος που δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Θα δούμε μέχρι το τέλος της μέρας αν κάποιος άλλος θα τον αντικαταστήσει από τους σοσιαλιστές ή αν θα το αναβάλουμε για άλλη φορά. Σημείο 2. Η έγκριση των πρακτικών της 6 Φεβρουαρίου του 2012. Δεν υπάρξουν παρατηρήσει. εγκρίνονται τα πρακτικά. Η σημερινή συνεδρίαση, συνάδελφοι, όπως συχνά συμβαίνει, θα μεταδίδεται στο, από το web stream και να θυμίσω επίσης στους συναδέλφους ότι απόψε για να εορτάσουμε την 50η επέτειο της κοινή γεωργικής πολιτικής εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο στις 7.30 το βράδυ θα κάνουμε μια δεξίωση, ένα κοκτέιλ μαζί με τους Υπουργούς Γεωργίας. Πάρα πολλοί Υπουργοί ήδη έχουν πει ότι θα συμμετέχουν και γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να έρθετε κι εσείς γιατί είναι εξαίρετη ευκαιρία για άτυπες ανταλλαγές απόψεων ανάμεσα στους βουλευτές της Επιτροπής μας και τους Υπουργούς του Συμβουλίου Γεωργίας. Αυτό θα γίνει απόψε στις 7.30. Και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα το εργαστήριο όσον αφορά τα αγαθά, τα κοινά αγαθά μέσα στη νέα κοινή γεωργική πολιτική, αντίκτυπος του πρασινίσματος και άλλε πιθανέ εναλλακτικέ λύσεις. Ενδιαφέρον το θέμα, να καλωσορίσω αμέσως τον αγαπητό Άλαν Μάθιους από το Trinity College του Δουβλίνου που θα μας παρουσιάσει την αξιολόγησή του για τις προτάσεις πρασινίσματος και όπως ήθεστε θα απαντήσει και στα ερωτήματα των συναδέλφων που θα θελήσουν να πάρουν το λόγο. Να χαιρετήσω τον εκπρόσωπο Μπάσκου της Επιτροπής και να δώσω αμέσως το λόγο στον φίλο και συνάδελφο Άλαν Μάθιους για την ε, εισήγησή του. Uh, <coughs> uh, Καλησπέρα σας και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα θερμά σας λόγια και για την πρόσκληση να ετοιμάσουμε αυτή τη μελέτη για την Επιτροπή για τα περιβαλλοντικά ε, δημόσια αγαθά και την ε, κοινή πολιτική. Θα ακούσετε βέβαια και την ε, οικονομική προοπτική απόψε. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε υπόψη πάντοτε ότι πρέπει να ακούσουμε και αυτούς που εργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της φύσης τη δηλαδή των περιβαλλοντικών αγαθών, διότι πρέπει πάντοτε οτιδήποτε κάνουμε να στηρίζεται στην βέλτιστη ε, επιστημονική γνώση και τις συμβουλές. Ελπίζω με την παρουσίασή μου να μπορέσω να σας πείσω για τις προτάσεις μας. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να ενισχυθεί η ε, ανταπόκριση με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τους θα ανταποκριθούν στους περιβαλλοντικούς, ε, στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχουμε θέματα όπως η βιοπικιλότητα, όπως ε, η, τα ύδατα, τα κλιματικές αλλαγές, τα διάφορα ε, ζυζάνια και ασθένειες η απώλεια οικοσυστημάτων, μάλλον υπηρεσιών οικοσυστήματος και η διάβρωση των εδαφών. Έτσι λοιπόν μπορούμε είτε να αγνοήσουμε είτε να αναβάλουμε δράση για, την περιβαλλον... για το πρασίνισμα της πολιτικής όπως ορισμένοι προτείνουν γιατί θα πρέπει να δοθεί λένε έμφαση στα τρόφιμα. Στην παραγωγή τροφιμών όμως το επιχείρημα αυτό δεν είναι καθόλου πιστικό για διάφορους λόγους. Καταρχάς διότι δεν έχω δει καμία μελέτη μέχρι τώρα η οποία να ε, στηρίζει τις ε, προτάσεις αυτές με προοπτική την παραγωγή των τροφίμων. Δηλαδή φαίνεται ότι από το, εάν εγκαταληφθεί το πρασίνισμα της πολιτικής της ΚΑΠ για να προωθηθεί η παραγωγή τροφίμων, πολύ μικρή διαφορά θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε 2% μόνο για την ζωική παραγωγή στο 2020 με 4% ε, χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τη βασική παραγωγή. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν λίγο πολύ την τάξη μεγέθος ε, της ανάπτυξης και της πτυτικότητας μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε κάθε χρόνο. Επιπλέον, η παραγωγή τροφίμων και η περιβαλλοντική υγεία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και όχι ως υποκατάστατα. Και τρίτον, η οσδήποτε ανησυχεί για την ποικιλία των γεωργικών πηγών πέραν της παραγωγής τροφίμων, θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να ε, κοιτάξει να καταργήσει την παραγωγή βιοκαυσίμων που είναι και πιο δαπανηρά και πολύ λιγότερο αιτιολογημένα ως παραγωγή όταν επιδιώκουμε την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Έτσι λοιπόν οι τιμές όταν είναι υψηλές μάλλον θα διατηρηθούν ψηλές ενώ το κόστος για την απώλεια, το, κόστος, το κόστος από την απώλεια των περιβαλλοντικών υπηρεσιών επίσης θα είναι πάρα πολύ υψηλό. Και επίσης μπορούμε να ε, αναλογιστούμε ότι όταν δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη των γεωργικών εισοδημάτων επιπλέον θα υπάρχει επιβάρυνση από την απώλεια οικοσυστημάτων. Και επίσης έχουμε και την ε, αβάσιμη ε, θεώρηση, το αβάσιμο αξίωμα ότι μπορεί το αποτέλεσμα του πρασινίσματος, μάλλον του προόδου προς την παραγωγή τροφίμων, να είναι οικονομικά ε, ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε πρέπει να προχωρήσουμε προς το πρασίνισμα της ΚΑΠΑ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τον πιο οικονομικό τρόπο για να το κάνουμε αυτό. Και έτσι περνάμε στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση τα εφιστάμενα μέσα που προσφέρει η κοινή γεωργική πολιτική και που είναι πρόσφορα για, την, για το πρασίνισμα. Δηλαδή η διασταυρώμενη ε, συμμόρφωση, και τα πολυετή προγράμματα. Και βέβαια ε, το check-up έδειξε ότι για πρώτη φορά μπορεί στον πρώτο πυλώνα να έχουμε καλά αποτελέσματα. Στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα λοιπόν, στο δεύτερο πυλώνα, έχουμε 4% αυτή τη στιγμή των, ε, των εδαφών, των εκτάσεων που μπορούν να υπαχθούν ανάλογα με το ρυθμό του προγράμματος, την περίοδο, το ποσοστό της χρηματοδότησης. Η συμμετοχή λοιπόν στη γεωργικά παύλα περιβαλλοντικά μέτρα προέρχεται από περιοχές ιδιαίτερως χαμηλής γεωργικής εκμετάλλευσης, χαμηλής έντασης γεωργικής εκμετάλλευσης ή από άλλες περιοχές όπου είναι υψηλότερο το κόστος της εκμετάλλευσης και άρα το, η συμμετοχή σε ένα αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα είναι πιο συμφέρουσα. Αυτό εξηγεί μια ποικιλία στη διαμόρφωση των αιτήσεων για συμμετοχή που οδηγεί βέβαια και στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προτάσεις οι ίδιες είναι γνωστές πιστεύω εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να δαπανίσω χρόνο για να τις ε, αναπτύξω, να σας τις υπενθυμίσω σημαντικό στοιχείο και ιδιαίτερα ως προς την δομή της κοινή γεωργικής πολιτικής, το πιο σημαντικό τμήμα δηλαδή του συνολικού νομοθετικού πακέτου και σημαντικό στοιχείο, είναι η ενίσχυση της όλης περιβαλλοντικής, των όλων περιβαλλοντικών επιδόσεων της κοινή γεωργικής πολιτικής μέσω του πρασινίσματος, μέσω συγκεκριμένων γεωργικών πολιτικών που θα αποβαίνουν εις όφελος του περιβάλλοντος και της γεωργίας και που θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούν όλοι οι γεωργοί. Και βέβαια 30% των αιτήσεων των ορίων για τα κράτη-μέλη θα αφορούν πλέον, θα προβλέπονται πλέον στην ε, κάλυψη των αναγκών εκείνων των γεωργών που τηρούν. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι γνωστά αυτά τα μέτρα, αυτές οι προτάσεις ε, προς το παρόν για να προχωρήσω σε σχόλιο για το καινούριο στοιχείο, για τα καινούρια στοιχεία της προτάσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, γιατί επιλέγει τη συγκεκριμένη προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιδίωξή της για το πρασίνισμα. Όπως είπα, ένα από τα θέλγητρα αυτής της επιλογής είναι ότι θα έχει οικουμενικό χαρακτήρα, δηλαδή θα πρέπει να ε, συμμετάσχουν σε αυτό όλοι οι παραγωγοί ε, σε αντίθεση με τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα τα οποία αφορούν ορισμένους μόνο. Δεύτερον, η έννοια της ορατότητας που είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράσινε πληρωμέ στον πρώτο πυλώνα θα μπορούν να νομιμοποιήσουν δηλαδή αυτέ τι πληρωμέ. Και επίση νόημα έχει και ω προ την πολιτική στήριξη, γιατί δεν υπάρχει πλέον πολιτική στήριξη για να συνεχιστεί η αυξημένη, ενισχυμένη, οι ενισχυμένε πληρωμέ για τον πυλώνα 2 που ξεκίνησε από το 2000 και έφτασε μέχρι το check-up πριν από μερικά χρόνια. Θα κοιτάξουμε τώρα τους λόγους ε, παράλληλα με τις προτάσεις. Το γιατί δηλαδή των μέτρων. Αλλά να δούμε και το πώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέτρων τα οποία ε, πληρούν τα εξής ε, τρία χαρακτηριστικά, τα οποία υποτίθεται πως είναι και απλά Ίσως αντίθετα από τα προγράμματα στον δεύτερο πυλώνα που θα είναι ίσως πιο στοχευμένα μένα αλλά με υψηλότερα ποσά και περισσότερο ε, ο κόστος. Δεύ, πρώτος, ε, πρώτος τρόπος. Δεύτερο πρέπει να είναι γενικευμένα, δηλαδή πρέπει να είναι δυνατόν να εφαρμόσετε σε, ολόκληρες, σε όλες τις εκτάσεις, σε όλων των εκτάσεων των γεωργικών σε όλα τα κράτη-μέλη, τα 27 δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ομοιογενή μέτρα απλά στην εφαρμογή τους και βέβαια τρίτον με ετήσιο χαρακτήρα, γιατί πρέπει να είναι και εκτελεστά και επαληθευτά, επαληθεύσιμα μάλλον, μέσα σε κάθε ετήσια ε, χρήση. Επίσης, μπορούμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες αν θέλετε στις επόμενες διαφάνειες, αλλά θα ήθελα καταρχάς να δώσω κάποιες ενδείξεις για αρχικές αντιδράσεις στις προτάσεις αυτές. Αντιδράσεις εκ των οποίων η μία ήταν παραδείγματι η επισήμανση αμφισημίας στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ότι ε, τέθη το ερώτημα αν πράγματι είναι δεσμευτικά τα μέτρα αυτά για τους, υποχρεωτικά δηλαδή για τους γεωργούς. Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον όρο mandatory, υποχρεωτικός. Προφανώς κάθε γεωργός έχει το δικαίωμα να μην ε, ενεργοποιήσει δικαιώματα ή απαιτήσει που μπορεί να έχει. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικά σε αυτό το βαθμό, αλλά από την άλλη ξέρουμε πώς λειτουργούν και οι πληρωμές με στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υποχρεωτικό μέτρο σημαίνει ότι ισχύει και για τον Γεωργό, ο οποίος δεν λαμβάνει ότι και τη βασική πληρωμή, την πράσινη πληρωμή, παρά μόνο εφόσον τηρεί τι ε, προποθέσει για το πρασίνισμα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή μια ερμηνεία περισσότερο των προτάσεων αυτών. Άρα θα έχουμε μια υπέρ διασταυρούμενη συμμόρφωση, δηλαδή θα υπάρχει διασταυρούμενη συμμόρφωση, η πολλαπλή συμμόρφωση, με τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και με τα τρία επιπλέον μέτρα πρασινίσματος. Εάν δοθεί αυτή η ερμηνεία λοιπόν στις προτάσεις, Στήσετε το ερώτημα γιατί να υπάρχουν δύο διαφορετικέ πληρωμέ με τη διαφορετική διαδικασία, τα διαφορετικά συστήματα, όλα αυτά, τα οποία βεβαίω περιπλέκουν όλη την κατάσταση. Άλλη ερμηνεία θα μπορούσε να είναι ότι η πράσινη πληρωμή είναι μια πληρωμή τύπου opt-in, δηλαδή εθελούσε συμμετοχή, όπου μπορεί ο κάθε γεωργό να αποφασίσει μόνο του ότι θέλει να συμμετάσχει και ω εκ τούτου αναλαμβάνει και του όρου αναλαμβάνει να τηρήσει τους όρους που συνδέονται με αυτό. Και άρα πλησιάζουμε σε ένα ρηχό θα έλεγα αγροπεριβαλλοντικό ε, μέτρο του πυλώνα 2 με συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον γεωργό περιορισμένες και βέβαια τη σχετική πληρωμή. Αν όμω δοθεί αυτή η ερμηνεία τότε καταλήγουμε στο ερώτημα γιατί να υπαχθεί στον πυλώνα 1 γιατί να να μην υπάγεται στον πυλώνα 2. Οι δύο επιλογές λοιπόν, είτε πιο αυστηρή δηλαδή ε, πολλαπλή συμμόρφωση ή περισσότερη έμφαση στην ενίσχυση των μέτρων του πυλώνα 2, θα είναι δύο εναλλακτικέ με τις οποίες θα βρεθούμε αντιμέτωποι κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης. Έχετε αντίγραφα του σχεδίου εκθέσεως. Θα επιτρέψτε μου λοιπόν να πω δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθώ να αναπτύξω την επιχειρηματολογία μου στηριζόμενο σε τρεις φάσεις. Η μία έχει να κάνει με την εξέταση των προτάσεων για πρασίνισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτόνομα, δηλαδή απλώς κοιτάμε εφόσον εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Μπορούν να τροποποιηθούν μπορούν ε, να βελτιωθούν, να ενισχυθεί το περιβαλλοντικό, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος ή μπορεί αντιθέτως ε, να οδηγήσουν σε κάποιες αναπάντεχες και αντίξωες συνέπειες. Δεύτερο στάδιο, προσπαθούμε να κοιτάξουμε με τη διεύρυνση του προγράμματος της ατζέντα δηλαδή. Μένουμε στα μέτρα του πυλώνα 1, αλλά με συμπληρωματικό ερώτημα εάν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει άλλου τύπου μέτρα που θα εφαρμόζονται μέσω του πρώτου πυλώνα και που ενδεχομένω, ιδιαίτερω μάλιστα, θα προσέφεραν περισσότερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Άρα, κοιτούμε την προοπτική τη μεγαλύτερη ευελιξία μέσα από τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ρίση όμω του πλαισίου, ημένοντα πάντα μέσα στο πλαίσιο του πυλώνα 1. Και στο τρίτο στάδιο διευρύνουμε ακόμη περισσότερο το πλαίσιο και λέμε ότι ναι, αν θέλουμε πρασίνισμα ακόμη περισσότερο, και αυτό γίνεται ήδη χάρη στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του πυλώνα 2, τότε να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε τον πυλώνα 2. Ίσως διασυνδέοντάς τον με τον πυλώνα 1 ή, εν πάση περιπτώσει, πάντως ε, δίνοντας περισσότερη έμφαση στα μέτρα αυτά του πυλώνα 2, τα αγροπεριβαλλοντικά. Αυτά είναι τα τρία στάδια της ανάλυσης, πάνω στα οποία στηρίζεται η ανάλυση. είναι και, αυτό είναι και το περίγραμμα της παρουσίασής μου. Και έτσι Ξεκινάμε με το πρώτο βήμα των ε, τριών προτάσεων της Επιτροπής και τους οικολογικούς χώρους ε, εστίασης που θεωρώ ότι μπορεί να θεωρούνται ως οι πιο περιβαλλοντικά πρόσφοροι από τους περισσότερους. Η Επιτροπή λοιπόν προτείνει 7% τουλάχιστον ε, των ε, επιλέξιμων νεκταρίων ενός ε, γεωργού, πέραν βέβαια των μονίμων βοσκοτόπων, να χαρακτηρίζεται ως χώρος οικολογικής εστίασης και δίνεται το σχετικό παράδειγμα του τι εννοείται με αυτό και στην αξιολόγηση συνεπειών ή αντικτύπου που δεν παρακολουθεί επακριβώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τον κανονισμό, δηλαδή κοιτάζει άλλα μέτρα όπως αυτό της ε, αγρανάπαυσης Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, ως προς την ε, χρήση αυτού του μηχανισμού αξιολόγησης που είναι η μελέτη αντικτύπου ως, ε, ως κριτήριο για την επιτυχία αυτού του συστήματος του, οικολογικού, του χώρου οικολογικής εστίασης. Εν πάση περιπτώσει όμως θα οδηγούσε σε ένα 5% χώρων οικολογικής εστίασης για 46% των γεωργικών γεών. Αυτές οι περιοχές λοιπόν, οι χώροι οικολογικής εστίασης, μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα και την πολυπικιλία επί παραδείγματι, πολυπικιλότητα, αλλά και φερρυπίν σε περίπτωση όπου ε, δημόσια γη χαρακτηρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο κοντά σε ε, υδάτινες πηγές, μπορεί να βοηθηθούν και οι υδάτινες πηγές. Και επίσης πολύ σημαντικό θα ήταν, ε, ξεκινώντας αυτή την παρουσίαση, να εξηγήσουμε ε, κατά πόσο αυτές τα περιβαλλοντικά αυτά ωφέλη από το σύστημα EFA, Ecological Focus Areas, μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε χωριστά γεωργική εκμετάλλευση ή θα πρέπει να έχει μια πιο εστιασμένη προσέγγιση. Και από αυτή την έννοια Δεχόμαστε ότι κάποιες εκτάσεις μπορεί να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα από την παραγωγή τροφίμων και άρα θα πρέπει να αξιοποιηθούν ως, ως εκτάσεις για παραγωγή τροφίμων, ενώ κάποιες άλλες λιγότερο ενδεχομένω. Και άρα η αχρανάπαυση θα μπορούσε να αφορά γες λιγότερο πρόσφαρες για, γεωργική, για παραγωγή τροφίμων. Δεν ε, είμαι ειδικό στην οικολογία. Νομίζω ότι εδώ όμω θα πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη και των επιστημόνων. Πάντως, έτσι κι αλλιώς ως θα έλεγε κανείς ότι εφόσον τα περιβαλλοντικά αυτά πλεονεκτήματα είναι απτά, εφόσον δηλαδή μπορούμε να αντικαταστήσουμε ε, κάποια κομμάτια γης χρησιμοποιώντας αυτή τη θεωρία, να περάσουμε δηλαδή σε άλλου χώρου, να περάσουμε σε άλλου χώρου την παραγωγή αυτή, ίσω θα μπορούσαμε έτσι πιο εύκολα να πετύχουμε το στόχο μα. Πάντως επειδή πολλά από τα θέματα τα οποία θα εξετάσουμε έχουν ω στόχο μια πιο απτή συγκεκριμένη προσέγγιση, γι' αυτό πρέπει να δούμε και θέματα δικαιοσύνη, διοικητικά, δικαιοσύνη δηλαδή μεταξύ των ίδιων των γεωργών, μεταξύ περιοχών, αλλά και τη σχέση κόστου και ε, ένα άλλο θέμα, προκειμένου να υποφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο, έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες. Ε, ποιες, ε, ποιους χώρους βάζουμε σε αγρανάπαυση, το 5%, το 7% που βρίσκονται οι περιοχές αυτές επί η υγεία αυτή, που βρίσκονται στο κέντρο ε, της αγροτικής περιοχής, στην άκρη της αγροτικής περιοχής, θα επιτρέψουμε ε, κάποια παραγωγή χαμηλής ε, έντασης, για παραγωγή τροφίμων, για παράδειγμα. Ή έπειτα θα υπάρχει σύνδεση μεταξύ των περιοχών αυτών, θα υπάρχουν κάποιοι διάδρομοι μέσα στο τοπίο ή θα είναι νησίδες. και επίσης να ξέρουμε κατά πόσο οι γεωργοί έχουν και τις συμβουλές που χρειάζονται έτσι ώστε να αποφεληθούμε περιβαλλοντικά όσο γίνεται περισσότερο. Άρα λοιπόν στις ζώνες ε, αυτές υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εκτός από την αγρανάπαυση αυτή καθεαυτή για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Έπειτα και ποια θα είναι η επίδρασή τους πάνω στην παραγωγή. Και αυτό θα ε, εξαρτηθεί από τη φύση της γης, από το σημείο που βρίσκεται η γη αυτή κλπ. κλπ. Τώρα, κάποια από τα θέματα τα οποία προέκυψαν στη συζήτηση για τις ζώνες αυτές, τα EFAs, έχει να κάνει με το μέγεθος των περιοχών πρώτα απ' όλα. Γιατί βάζουμε 7%, μήπως θα πρέπει να είναι περισσότερο, μήπως θα πρέπει να είναι λιγότερο. Η Επιτροπή στηρίζει το 7% στη βάση ότι πιστεύετε ότι έτσι επιτυχάνεται καλή ισορροπία. Δηλαδή έχουμε επαρκείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από την άλλη μεριά δεν έχουμε ε, κακές επιπτώσεις. Τώρα, ποια είναι η περιοχή βάσης για αυτό το 7% ή για όποιο ποσοστό πάνω στο οποίο τελικά θα συμφωνήσουμε, αυτό έχει να κάνει με τα προσωρινά βοσκοτόπια, με ε, την, τις καλλιέργειες. Έπειτα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και το διοικητικό σκέλος. Μερικές φορές δηλαδή δυσκολευόμαστε γιατί δεν ξέρουμε τι στοιχεία πρέπει να συμπεριλάβουμε μέσα σε αυτά που ζητάμε από τους γεωργούς. Υπάρχουν στοιχεία πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Το θέμα δεν είναι μόνο το αν υπάρχει κάπου ένας φράχτης, πρέπει να ξέρουμε. Υπάρχει ας πούμε ένα δέντρο στη μέση του αγροτεμαχίου και είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο χρειαζόμαστε για να καθορίσουμε τις ζώνες αυτές. Οι αγρότες πρέπει να τις ξέρουν αυτές τις ε, λεπτομέρειες και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο μέσα στον κανονισμό αλλά και στις εφαρμοστικές πράξεις. Θα επανέλθω σε αυτό για το κατά πόσο τα EFAs πρέπει να είναι οικουμενική απέτηση ή όχι. Μήπως πρέπει τις περιοχές αυτές να τις συνδέσουμε με την αγρανάπαυση. Αν για παράδειγμα σε μια περιοχή έχουμε πολλά δάση, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες ζώνες είναι μικρή. Ενώ αν έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο τα πράγματα αλλάζουν. Έπειτα, πώς θα έχουμε τη βιοπικιλότητα καλύτερα. Μπορούμε να σκεφτούμε και το θέμα της ε, εμπορίας οικολογικών ε, τέτοιων περιοχών. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπρεπε παντού να υπάρχει αυτό το 7%, αλλά σε περιοχές όπου αυτό κοστίζει περισσότερο, οι αγρότες θα μπορούσαν εντό αγωγικών να αγοράσουν ε, ένα ποσοστό από αγρότες οι οποίοι δυσκολεύονται λιγότερο να βάλουν σε αγρανάπαυση τη δικιά τους γη. Όλα εξαρτώνται βέβαια και από αυτά που θα πούν οι ειδικοί επί της οικολογίας, προκειμένου να πετύχουμε την βιοπικιλότητα και άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. Έπειτα, πώς ενθαρρύνουμε την κατάλληλη διαχείριση των οικολογικών αυτών περιοχών. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ε, ελάχιστα κίνητρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η γη η οποία βρίσκεται σε αγρανάπαυση για τέτοιους ε, λόγους. Υπάρχουν παραδείγματα και δυνατότητες οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό σημείωμα. Ορισμένοι θα πούν ότι πρέπει να εφαρμόσουμε και σε αγροτικές περιοχές, γενικά τις οικολογικές αυτές ε, περιοχές, αλλά και γενικότερα σε αγροτικές περιοχές γενικότερα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στην πράξη είναι αναπόφευκτο να υπάρχει κάποια ελαστικότητα στο σύστημα. Ξέρουμε ότι πολλές αγροτικές ιδιοκτησίες δεν είναι ενιαίες, είναι κατακαιρματισμένες. Οπότε ακόμα κι αν μια εντατική καλλιέργεια αποφασίσει να νοικιάσει, ο ιδιοκτήτης δηλαδή να νοικιάσει ένα κομμάτι σε κάποια άλλη περιοχή που είναι λιγότερο παραγωγική από πλευρά τροφίμων, πώς θα το εξετάσουμε αυτό. Πώς θα το θεωρήσουμε, θα το θεωρήσουμε ένα παραθυράκι ή θα θεωρήσουμε ότι απλώς επιτρέπει μια ελαστικότητα στο σύστημα. Και άρα θα το δούμε με καλό μάτι. Τώρα, μια άλλη πρόταση της Επιτροπής είναι η διαφοροποίηση των καλλιεργών, καλλιεργιών. Εκεί όπου η αρρώσιμη γη ενός αγρότη καλύπτει πάνω από τρία εκτάρια και δεν χρησιμοποιείται πλήρως ως ε, σκοτόπιο, πάντα δεν καλλιεργείται, η καλλιέργεια στην αρρώσιμη γη θα πρέπει να έχει κάποια νότοτα και κάποια ελάχιστα ποσοστά. Η διαφοροποίηση αυτή προσφέρει πλεονεκτήματα στο περιβάλλον. Για παράδειγμα γίνεται χαμηλότερη εκμετάλλευση, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι επιθυμητό. Αλλά αυτό καθορίζεται διοικητικά κανονικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση αντικτύπου λέει ότι το μέτρο αυτό θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο, γιατί μόνο ένα 3% της αρρώσιμης γης θα επηρεαστεί. Ενώ αλλού το κόστος θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Άλλες μελέτες τώρα που έχουν κάνει τα κράτη-μέλη λένε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερος αντίκτυπο σε περισσότερα αγροτεμάχια από μια τέτοια πρόταση. Οι επιπτώσεις πάντως εξαρτώνται και από το πώς ορίζεται η εισοδιά. Ε, πρόκειται για μόνιμες καλλιέργειες, για παράδειγμα για μπέλια. Έπειτα αν, υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει αγροτική γη με μεικτή κτηνοτροφία. όπου καλλιεργούνται και ζωοτροφές για παράδειγμα. Τι θα πούμε, θα πούμε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές σοδιές, Οπότε το κίνητρο μπορεί να είναι να βγει από την ρώσιμη παραγωγή και να έχει μόνο βόσκο τόπια. Οπότε τότε έχουμε ε, μόνο καλλιέργεια και είναι ακριβώς το αντίθετο από τη διαφοροποίηση που θέλουμε. Έπειτα το όριο των τριών εκταρίων μήπως θα πρέπει να αυξηθεί και να ασχοληθούμε περισσότερο με το 70% όριο το οποίο ενδεχομένως μπορούσαμε να το αυξήσουμε στο 85%. Το τρίτο μέτρο είναι να παραμείνουν ε, τα μόνιμα βοσκοτόπια. Οι αγρότες ε, σκέφτονται εν ώψη του 2014. Εδώ όμως είναι ένα διαφορετικό μέτρο, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ήδη κάποια διάταξη στον κανονισμό για τις άμεσες πληρωμές που λέει ότι το κράτος μέλος πρέπει να διαβεβαιώσει ότι το ποσοστό γης που βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμου σκοτοπίου πρέπει να είναι συγκεκριμένη σε σχέση με το συνολικό και δεν θα πρέπει να απομακρύνεται από το 10%. Η πρόταση της Επιτροπής ε, λοιπόν αυτό τον περιορισμό που υπάρχει σε εθνικό επίπεδο θέλει να τον γενικεύσει σε επίπεδο αγροτικής γης. Τώρα έχει νόημα ή όχι. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο στόχος μας τι είναι, είναι οι κλιματικές αλλαγές, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, δηλαδή πώς θα αποφύγουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ή είναι η ενίσχυση της διαφοροποίησης των καλλιεργών. Γιατί εδώ δεν επικεντρώμαστε τελικά σε περιοχές με συγκεκριμένη φύση καλλιέργειας, Τώρα θέματα εδώ πέρα, ελαστικότητας ή διοικητικών προβλημάτων ή κατά πόσο το έτος 2014 αναφοράς είναι κάτι καλό ή όχι. Αυτά είναι λεπτομέρειες που έχουν ε, τεθεί ήδη σε κάθε συζήτηση που γίνεται για αυτό το θέμα. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο στάδιο. Είδαμε τα τρία μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα αναρωτιόμαστε υπάρχουν άλλα ενδυνάμει μέτρα ή άλλα στοιχεία ευκαμψίας, ελαστικότητας για το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα. Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς τι θα μπορούσε να είναι, εφόσον θέλουμε να είναι κάτι απλό, γενικευμένο και τίσιο. Η περιτροπής ε, σοδιά είναι κάτι είναι μια οικολογική απέτηση έτσι κι αλλιώς για την πληρωμή ε, των αγρότων. Επίσης για ένα υψηλό ποσοστό βοσκοτόπων και αυτό υπάρχει σε κάποιο άλλο μέτρο. Άλλες ιδέες όμως που ακούγονται είναι ιδέες που δεν θυμίζουν τόσο πολύ μέτρα πρώτου πυλώνα. μέτρα πράσινη ανάπτυξη, για παράδειγμα βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τεθούν σε εφαρμογή στον πυλώνα 1. Έπειτα ερχόμαστε στο ενδιαφέρον θέμα που λέει αν θέλουμε να έχουμε ένα μέτρο για όλους δεν θα έπρεπε να προσφέρουμε περισσότερη ελαστικότητα στα κράτη-μέλη τότε για τα πράσινα μέτρα τα οποία αποφασίζουν να υιοθετήσουν. Έχουμε την προσέγγιση που μιλάει για ένα μενού, έχουμε την προσέγγιση βάση του γκάικ και έχουμε και το green by definition και αυτή την προσέγγιση, δηλαδή εξορισμού πρασίνισμα. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε το μενού και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν. Η αναλλακτική ποια είναι, είναι ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να αποφασίσουν για ένα πακέτο μέτρου από μία λίστα και μετά οι αγρότες να αποφασίζουν ανάμεσα στα μέτρα αυτά. Βέβαια το πρόβλημά μου με το πρώτο είναι ότι είναι δύσκολο να φανταστούμε επιπλέον απλά μέτρα για τον πυλώνα 1 από τα οποία να μπορούν να διαλέξουν τα κράτη-μέλη. Οπότε τελικά μιλάμε για ελαστικότητα σε επίπεδο του αγρότη όταν μιλάμε για το μενού. Και όπως είπα, πολλές από τις προτάσεις που είναι εδώ μου φαίνονται ότι καλύπτονται περισσότερο από τον πυλώνα 2 παρά από τον πυλώνα 1. Ένας τρόπος πάντως ελαστικότητας που μπορούμε να έχουμε σε επίπεδο αγροτών είναι η εξαίρεση του green by definition. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Στην πρόταση αυτή της Επιτροπής που λέει ότι οι βιολογικές καλλιέργειες ήδη συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του πυλώνα 1, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα παραπάνω και μπορούν να κρατήσουν ό,τι πληρωμές παίρνουν από τον πυλώνα 2. Βέβαια τα κράτη-μέλη μπορούν να πούν γιατί μόνο οι καλλιέργειες, γιατί όχι και άλλες καλλιέργειες οι οποίες εντάσσονται σε προγράμματα αγροπεριβαλλοντικά και καλύπτουν ε, κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μήπως θα έπρεπε να ξερούνται επίσης από τις απαιτήσει συμμόρφωσης. Εγώ νομίζω ότι αυτό βέβαια θέτει το θέμα της διπλής χρηματοδότησης. Δηλαδή τελικά οι αγρότες θα πληρώνονται δύο φορές για την ίδια πρακτική που ακολουθούν. Και θέτει και το ζήτημα που λέει ότι αν κάνουμε μια μεγάλη εξαίρεση για κάποιους αγρότες που ήδη συμπεριλαμβάνονται σε τέτοιου είδου προγράμματα, τότε τι επιπλέον όφελος έχουμε για το περιβάλλον και για τον καταναλωτή. Ένας άλλος τρόπος για να πετύχουμε την ελαστικότητα στον πυλώνα 1 είναι μέσω των ε, ήδη υπαρχουσών ε, προδιαγραφών για την καλή διαχείριση. Η Κομισιόν δεν το κοίταξε αυτό. Το απέρριψε λέγοντας ότι δεν προσφέρει μια οικομενική εφαρμογή από τα κράτη μέλη, ότι τα κράτη-μέλη δηλαδή ερμηνεύουν διαφορετικά τις προδιαγραφές αυτές. Δεν θα υπήρχε επίσης επαρκής προβολή ε, του μέτρου με τις ε, πληρωμές, δηλαδή περισσότερο θα επικεντρωνόμαστε στην πληρωμή και όχι στον τρόπο με τον οποίο επιτυχάνεται η πληρωμή και ότι θα υπήρχε μεγάλη αντίσταση από τους αγρότες που θα θεωρούσαν ότι τους επιβάλλεται ένα μέτρο. Όμως δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχουν θετικά στοιχεία. Τα κράτη-μέλη έτσι κι αλλιώς ε, είναι εξοικειωμένα με διπλές προδιαγραφές. Είναι σωστό τα δι... τις διπλές αυτές προδιαγραφές να τις ερμηνεύουμε διαφορετικά ανάλογα στο... σε ποιο κράτος είμαστε. Έπειτα, για να υπάρχει πολιτική προβολή, το θέμα είναι να ξέρουμε κατά πόσο υπάρχουν περιβαλλοντικά κέρδη. Τότε πολιτικά πρέπει να υπάρχει στήριξη μακροπρόθεσμα. Τώρα πριν φύγουμε από τον πυλώνα 1 πρέπει να υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το κόστος. Το 30% των άμεσων πληρωμών είναι κάτι που τίθεται υπό αμφισβήτηση. Γιατί 30, μήπως θα πρέπει να είναι 20, μήπως θα πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Και αν είναι σε θελοντική βάση, τότε τι γίνεται με τις πληρωμές οι οποίες τελικά δεν χρησιμοποιούνται. Τι επιπτώσεις η υπάρχουν στη, από τις ε, πράσινες πληρωμές στο ρυθμό με τον οποίο γίνονται αλλαγές. Το θέμα του ελέγχου και της ε, αξιολόγησης είναι θέμα στο οποίο δεν προλαβαίνω να μπω τώρα, αλλά αν έχετε ερωτήσεις ευχαρίστω να σας απαντήσω. Τέλος, επιτρέψτε μου να έρθω και στο τρίτο στάδιο και θα το κάνω αυτό πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Το πρασίνισμα μέσω του δεύτερου πυλώνα. Αυτό είναι όντως μια ελκυστική προσέγγιση. Θα μπορούσαμε να την ε, δούμε σοβαρό. Τα κράτη-μέλη είναι εξοικειωμένα εξάλλου με τα προγράμματα του πυλώνα 2. Η ένσταση εδώ είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εξίσου συμμετοχή από παντού, δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, κυρίως στην ε, στις εντατικές καλλιέργειες. Το πρασίνισμα βέβαια μέσω του πυλώνα 2 εξαρτάται και κατά πόσο θα αυξηθεί όχι ο προπολογισμό εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολιτικές αντιρρήσεις επ' αυτού. Εν κατακλείδη. Υπάρχουν διάφορες επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Εξαρτάται βέβαια αν θέλουμε να περιοριστούμε στις τρεις προτάσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε και τις επιλογές ελαστικότητας και κατά πόσο θέλουμε να ανοίξουμε το ζήτημα που λέει θέλουμε αποκλειστικά μέσω του πυλώνα 2 να πετύχουμε το πρασίνισμα ή περισσότερο μέσω του πυλώνα 2 από ό,τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκεπτόμενοι όλα αυτά, εγώ που καταλήγω. Καταλήγω στο ότι δεν υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση που να κυριαρχεί όλων των κριτηρίων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Αν θέλουμε ένα οικουμενικό μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται παντού σε όλε τι αγροτικέ εκμεταλλεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα έχουμε τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Άρα δεν θα έχουμε μεγάλα ωφέλη πρασινίσματο Και μπορούμε βέβαια να αναρωτηθούμε και κατά πόσο αξίζει τον κόπο. Αν βέβαια θέλουμε να έχουμε πιο στοχευμένα μέτρα, τότε αμέσως γίνεται πιο περίπλοκο γραφειοκρατικά το ζήτημα. Τίθεται το θέμα της δικαιοσύνης μεταξύ των χωρών μελών, πώς λέει θα αξιολογήσουμε μια χώρα κατά πόσο θα κάνει καλά τα πράγματα και πώς θα αξιολογήσουμε μια άλλη χώρα. Οπότε αυτό που έχω κάνει εγώ στην έκθεση είναι ότι προσπαθώ να δω από πού ξεκινάμε για να πάρουμε αποφάσεις, δηλαδή τι εναλλακτικέ είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Σίγουρα θα υπάρξουν και αυτοί που θα πούν ότι δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε το πρασίνισμα σε αυτό το στάδιο και η δικιά σας επιλογή είναι είτε να το ξεχάσουμε τελείως το στοιχείο αυτό του πρασινίσματος ή να αποδυναμώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ δεν θα σύστηνα μια τέτοια προσέγγιση, αλλά είναι μια εναλλακτική που υπάρχει κάποιος θα μπορούσε να στηρίξει την πρόταση της Επιτροπής ε, τροποποιώντας κάποια στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί στη συζήτηση. Έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε πράγματι. Μπορείτε να αποφασίσετε ότι πράγματι η ελαστικότητα είναι κάτι σημαντικό και είσαστε διατεθειμένοι να παζαρέψετε κάποια επιπλέον διοικητικά μέτρα και κάποια ερωτηματικά για την ε, ισοδυναμία μεταξύ των χωρών μελών, προκειμένου τελικά να έχετε πιο αποτελεσματικά περιβαλλοντικά μέτρα συνολικά. Ή μπορεί και να αποφασίσετε ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσετε να βρείτε περισσότερα χρήματα για τον πυλώνα 2 ή να χρησιμοποιήσετε περισσότερο τα χρήματα του πυλώνα 2 για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και έτσι να αποφασίσετε τελικά ποιο είναι ο πιο αποτελεσματικό και στοχευμένο τρόπος για να πετύχετε το πρασίνισμα. Πάντως επιπλέον κάποια οικουμενικά μέτρα όπως για παράδειγμα να αυξήσετε την ε, γραμμή, τη βασική, τη βάση σας δηλαδή, συμπεριλαμβάνοντας σιγά σιγά όλο και περισσότερες ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρόγραμμά σας. Έτσι ολοκληρώνω την παρουσίασή μου, Πρόεδρε, και βέβαια με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τις αντιδράσεις στην αίθουσα. Ευχαριστώ. Bene, grazie, grazie al Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ καθηγητά Άλαν Μάθιο, πολύ υλικό. Έχουμε ήδη πολλούς εγγεγραμμένους που έχουν ζητήσει το λόγο και γι' αυτό ξεκινάμε αμέσως με τον κύριο Λένετσεκ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι υπέρ μιας απόλυτα οικολογικής γεωργίας. Ανέκαθεν ήμουν υπέρ τέτοιου τύπου γεωργίας και θα εξακολουθήσω να είμαι υπέρμαχος ε, της οικολογικής γεωργίας. Νομίζω πως πρέπει ακόμα πολλά να γίνουν ώστε η γεωργική παραγωγή να σέβεται τους περιβαλλοντικούς κανόνες και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει ένα ε, επαρκή όγκο ε, τροφίμων χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον. Όταν όμως ακούω αυτή τη συζήτηση και αναλύω την ε, θέση της, ε, της προτάσεις μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η άποψή μου ότι ε, όλες αυτές οι προτάσεις που μας παρουσιάζει η Επιτροπή δεν ανταποκρίνονται καθόλου στις προσδοκίες μου. Εμείς Έχουμε πληρώσει εξαιρετικά ακριβά τη γεωργική πολιτική και όλες αυτές οι προτάσεις θα κοστίσουν και πολύ ακριβά και δεν προσφέρουν πραγματικά προστιθέμενη αξία. Στο μέλλον, για παράδειγμα, δεν θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Οι συνήθειες των γεωργών δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και ωστόσο, αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας Θα πρέπει επίση να αποδείξουμε ότι μπορεί κανείς να κερδίσει χρήματα κάνοντας πράσινη παραγωγή τροφίμων και οικολογική παραγωγή. Την ώρα αυτό δεν είναι δυνατόν. Ένας γεωργό που έχει 5-10 εκτάρια πώ μπορεί να πουλήσει με τα επιπλέον έσοδά του με βάση το δεύτερο πυλώνα. Σήμερα αυτό δεν είναι δυνατόν. Ακόμα και οι μεγάλοι ε, σε επιχειρήσεις σε άλλους τομείς, ε, ε, στο ορυχία, στον άνθρακα, οι χαλιβουργίες δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν σε μια ανταλλαγή ε, ποσοστώσεων για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Και τι να πει ένας μικρός ε, γεωργός. Εάν θέλουμε να εισάγουμε τέτοιου είδους στρατηγικές για τις μικρές εκμεταλλεύσεις στη γεωργία, νομίζω ότι πολύ θα κερδίσουν πολλά, αλλά όχι οι γεωργοί. Αναφέρεται το παράδειγμα της Ελβετίας. Είναι ένα πολύ ε, δυνατό παράδειγμα. Μπορούμε να αντιγράψουμε πολλά πρότυπα από τους Ελβετούς, αλλά όσον αφορά τη γεωργία πιστεύω πως θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφέρουμε τις δικούς τους κανόνες εδώ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα δεν είναι καν να καταστήσουμε άλλους τομείς ο, ο, ο τραπεζικός τομέας, ας πούμε, που είναι πολύ ισχυρός στην Ελβετία, ε, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το τραπεζικό σύστημα της Ένωσης. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι θα αντιγράφουμε ό,τι κάνουν οι Ελβετοί, ούτε μπορούμε να συγκρίνουμε. Είμαι λοιπόν αντίθετο σε αυτές τις ε, προτάσεις. Άκουσα μάλιστα επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία θα έπρεπε να εξετάσουμε κατά πόσο πρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε τρόφιμα ή αν θα πρέπει να παράγουμε μόνο φυτά για τα βιοκαύσιμα. Όταν ακούω τέτοιου είδου επιχειρήματα, πραγματικά ανησυχώ, γιατί για χρόνια προσπαθούσαμε να πείσουμε τους γεωργούς μας να καλλιεργούν περισσότερο για τα βιοκαύσιμα και τώρα μιλάμε για εναλλακτικέ. Θέλουμε να αλλάξουμε πορεία στην ουσία. Θέλουμε να εγκαταλείψουμε την παραγωγή βιοκαυσίμων, αλλά ταυτόχρονα να εισάγουμε νέους περιορισμούς. Αυτό θα σήμαινε ότι εγώ Περίμενα σήμερα η Κομισιό να μας παρουσιάσει συγκεκριμένους λογαριασμούς, δηλαδή ποιες είναι οι επενδύσεις για τα βιοκαύσιμα, ποιες είναι οι απώλειες που συνδέονται με το γεγονός ότι παράγουμε καλλιέργειες για τον τομέα των βιοκαυσίμων και όχι για την ε, ανθρώπινη κατανάλωση και ποια θα ήταν τα νέα στοιχεία με βάση τις νέες προτάσεις, αν βασιστούμε στις νέες προτάσεις, γιατί αυτά θα αλλάξουν κάπως, για παράδειγμα, τον τομέα της, ε, των παραγωγικών δυνατοτήτων. Με άλλα λόγια, έχω τεράστιες αμφιβολίες, κύριε Πρόεδρε. Από τη μια πλευρά είμαστε όλοι πεπισμένοι, νομίζω, αν εφεξαιρέσεις ότι ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Όμως ε, αμφιβάλλω γιατί αυτά τα μέτρα δεν είναι καν ε, υποχρεωτικά. Πράγμα που με κάνει να αμφιβάλλω πολύ. Νομίζω πως δεν ε, λειτουργούμε με βάση τις προσδοκίες ε, των ε, γεωργών, αλλά με, με βάση τα συμφέροντα που ισχύουν σήμερα. Πώς θα μπορέσουμε να βρούμε την ισορροπία Είπατε πως θα ήταν μια δίκαιη πρόταση, όμως οι γεωργοί στα περισσότερα κρατημέλη θα λάβουν ε, πληρωμές με διαφορετικά επίπεδα, γιατί 30% για τους γεωργούς στη Γαλλία δεν είναι το ίδιο ποσό σε απόλυτους όρους για έναν Γάλλο γεωργό όπως για έναν Ρουμάνο γεωργό, όμως η προσπάθεια θα είναι η ίδια. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες αφιβολίες, ανοιχτά ζητήματα. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να τα αποσαφηνίσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης και μάλιστα είμαι πολύ ικανοποιημένος που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα και μπορώ να συμμετέχω σε αυτή, αλλά επαναλαμβάνω έχω πολλές αμφιβολίες και θα σας τις δώσω και γραπτός κύριε Πρόεδρε, γιατί καταρχήν αυτό αφορά το κόστος, το κόστος διαχείρισης, το, τα κόστη που συνδέονται με τα διάφορες αυτές αλλαγές, όπως στον τομέα των βιοκαυσίμων για παράδειγμα, νέες προτάσεις για τους γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς, τον οποίο την παραγωγή περιορίζουμε, ενώ ταυτόχρονα εισάγουμε άλλες λύσεις που θα σημάνουν μεγαλύτερη χρήση ε, χημικών λοιπασμάτων και ούτω καθεξής. Με πολλές αμφιβολίες λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Σας ζητώ να κρατάτε το χρόνο ομιλίες γιατί είναι πολλοί οι που έχουν ζητήσει το λόγο. υπάρχουν ειδικά θέματα, Σα θυμίσω ότι πέρα από τον πρωτοκαθηγητή Άλαν Μάθιο, η δική μας υπηρεσία μπορεί να βοηθήσει. Ο Τζον Λάινερ. Πρόεδρε, πολύ σύντομο. Διαδικαστικό έχετε. Να ορίσετε μέγιστο χρόνο Τρία-τέσσερα λεπτά το πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τρία-τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σας κρατήσω λιγότερο ακόμα. Καταρχάς, ευχαριστώ τον καθηγητή Μάτθιους για την εξαιρετική παρουσίαση. Και επίσης, στο διάγραμμα που έχει ε, παρουσιάσει δίνει ακριβώς το νόημα όλων αυτών των προτάσεων. Και ιδιαίτερα μου φάνηκε ενδιαφέρουσα η συσχέτιση μεταξύ πρασινίσματος και προπολογισμού. Εάν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε από ό,τι φαίνεται και άλλες περικοπές στον συνολικό προπολογισμό του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από τα πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές, ε, θα ήταν καλό να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε στις προτάσεις της Επιτροπής προς τον προπολογισμό. Θα ήταν καλή δηλαδή ε, στρατηγικά μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη και αυτή, αυτό το ενδεχόμενο. και τον όγκο της ΚΑΠ. Επίσης, απλούστευση ή περίπλοκη δομή είναι μια λεπτή ισορροπία την οποία θα πρέπει να αναζητήσουμε. Πάντως, αν αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την κοινωνική πολιτική ε, για τη γεωργία, ασφαλώς δεν ξεκινάμε από το σημείο αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε από πού ξεκινάμε και πού τίνουμε με τις πολιτικές μας επιλογές. Δεν θέλω να τον καθηγητή Μάθιους. Εάν θεωρεί ότι στο πρασίνισμα η βιολογική παραγωγή αυτομάτως μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία αυτή. Γιατί εδώ δεν είναι σαφές ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Δηλαδή, καταρχάς ε, ανήκει στην ορολογία ή ε, στη, στους χαρακτηρισμούς του ΠΟΕ. Πρώτον και δεύτερον, διπλή χρηματοδότηση. Ένα ζήτημα στο οποίο η Επιτροπή, η Επιτροπή δεν μου έχουν δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί εφόσον η ιδεολογική παραγωγή υπάγεται στο πρασίνισμα αυτομάτως, τότε η Natura 2000 και η περιβαλλοντικά χαρακτηρισμένη γεωργική παραγωγή επίσης θα πρέπει να επαχθεί σε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να πιέζω, το ξέρω, αλλά θα ήθελα πιο συγκεκριμένε απαντήσει για το πώς, μπορούν, πώς μπορούμε να χειριστούμε τις προτάσεις της Επιτροπής ως προς τη συγκεκριμένη αυτή έννοια. Ευχαριστώ, Μάρτιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χόισλινγκ. Ευχαριστώ ιδιαίτερω για την παρουσίαση που πάντα, όπω μια κάθε καλή παρουσίαση, γεννά πιο πολλά ερωτηματικά από τι απαντήσει που δίνει. Τα βιοκαύσιμα βεβαίω είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στη συζήτηση. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αναδύεται σε πολλά κράτη-μέλη όπω τη Γερμανία ιδιαίτερω, που δεν μπορούμε φυσικά να το παραγνωρίζουμε, αλλά και η Ευρωπαϊκή Οδηγία θα επηρεάζει περισσότερο τα ιεραρχικά μας συστήματα από ό,τι θα θέλαμε ενδεχομένω. Και επίσης ε, μια πολιτική προσέγγιση ε, που προκύπτει μέσα από την κοινή γεωργική πολιτική δεν μπορεί να παραγνωρίσει αυτή τη διάσταση και την αιτιολόγηση των γεωργικών πληρωμών. Ένα σημαντικό σημείο λοιπόν και ερώτημα είναι εάν αρκούν τα μέτρα για μια βιώσιμη γεωργία. τότε όταν είχαμε ξεκινήσει είχαμε ε, ορίσει σαν βασική αρχή ότι για να επιδοτείται μια παραγωγή πρέπει να δίνει συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένο καρπό δηλαδή. Ε, τώρα έχουμε άλλες επιλογές και ίσως ε, χρειάζεται να δούμε την ε, αντιμετώπιση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, δηλαδή γεωργικές επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους με διαφορετική μεταχείριση να αντιμετωπίζονται από ότι μικρότερες. Έχουμε επίσης το ζήτημα των... Ε, των οσπρίων και όταν τα προβλήματα εμφανίζονται στις περιοχές μόνο της εντατικής καλλιέργειας, θα πρέπει να μεριμνήσουμε να είναι δεσμευτικά τα μέτρα για όλους, για εκείνους ιδιαίτερους που έχουν τα προβλήματα και να είμαι σε θέση να διαθέτουν απεριόριστα το πλεονάζον αυτό προϊόν στο οποίο καταλήγουν, έτσι ώστε να μεταθέτουν το πρόβλημά τους σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες δεν έχουν στην πραγματικότητα δυσκολίες. Ή θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν κατάλογο, ένα shopping list που να πούμε τι μπορούμε να έχουμε, τι δεν μπορούμε να έχουμε, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Όλα αυτά δεσμευτικά με απλούς όρους αναγνωρίσιμο για την κάθε περιοχή έκταση γεωργική εκμετάλλευση. Γιατί βεβαίω εάν ε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένε προδιαγραφέ και αν είναι εκούσια η συμμετοχή, τότε μπορεί και να ακυρωθεί το ίδιο το νόημα των μέτρων, διότι απλώς δεν θα εφαρμόζονται όπως πρέπει. Εδώ τεθεί και το ζήτημα του δεύτερου πυλώνα. Δεν είναι δεσμευτικός δεύτερος πυλώνας. Ή τότε δεν θα έπρεπε να περάσουμε από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα και να ισχύει ο δεύτερος πυλώνας ως υποχρεωτικός για κάθε εκμετάλλευση. Όπου όμως τίθεται το άλλο πρόβλημα, μεγάλο για ορισμένα κράτη-μέλη, αυτό της εγχρηματοδότησης. Γιατί στα μεγέθη που έχουμε τώρα, στα ποσοστά δηλαδή επί των εκτάσεων που προβλέπονται τώρα, ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να έχουν σημαντικέ δυσκολίε. Άρα μπορεί να είναι καλό ο σκοπό, αγαθό ο σκοπό, αλλά στην πράξη μπορεί να μην επαρκούν τα κονδύλια για την πραγματική υλοποίησή του, για την πρακτική υλοποίησή του. Χαίρομαι λοιπόν και καλωσορίζω την πολιτική προσέγγιση, την πολιτική επιλογή, αλλά ε, ενδέχεται να αντιμετωπίσει πάρα πολλέ επικρίσει. και ίσως θα έπρεπε να επανεξετάσουμε το ζήτημα του υποχρεωτικού ή μη χαρακτήρα των μέτρων. Ευχαριστώ, Άλμπερτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας άκουσα προσεκτικά, κύριε καθηγητά. Υπάρχουν κάποια σημεία από την παρέμβαση στα οποία μπορώ να ε, υποστηρίξω και εγώ ρητά, αλλά όπως και ο κύριος Χόισλινγκ, γεννούν μια σειρά από νέα ερωτηματικά. Και θεωρώ ότι όντω η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον ε, υλοποιηθεί, οι προτάσει, μάλλον είναι πολύ, πιο, πολύ περίπλοκες και μπορούν να οδηγήσουν περισσότερη γραφειοκρατία. Άρα οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραγνωρίζουν ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει στον χώρο τη γεωργική Πολιτική. Και βλέπουμε στην πρόταση Τη εκθέσεως που εγκρίθηκε με 90% ε, από το Κοινοβούλιο και στην πρώτη έκδοση τη έκδοση Lion, ότι επιδιώκεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λιγότερη γραφειοκρατία, ενώ το, το πρόγραμμα, οι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στείλουν προ το αντίθετο. Αυτό το οποίο πάντοτε με ενοχλεί είναι ότι έρχεται πάντα κάποιο να βρει νέα συστήματα, να εφεύρει νέα συστήματα. Μέτρα τα οποία δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί από ορισμένα κράτη-μέλη. Ε, εν πάση περιπτώσει, να σα πω τι συμβαίνει στην ε, Αυστρία την, την ε, Βαβαρία ή άλλα κράτη. Κοιτάξτε τι συμβαίνει εκεί όπου υπάρχει ε, λειτουργία του συστήματος υπό το δεύτερο πυλώνα με γεωργικά μέτρα που εφαρμόζουν ουσιαστικά τη δε... το δε Σάββατο που ήμουνα στο χωράφι μου, ανέβηκα στο τρακτέρ μου και ε, φρόντισα την καλλιέργεια της θερινής μου παραγωγής ε, που θα εξασφαλίσει επαρκή δίνη για την ζηθοποιία της Βαβαρίας το επόμενο φθινόπωρο. Έτσι λοιπόν... Δίπλα στο χωράφι μου έχει οριστεί ένας χώρος ε, πράσινος ο οποίος δεν, ασχολ, δεν καλλιεργείται από κανέναν, έχει να κάνει μόνο με όλους αυτούς τους ε, περιβαλλοντολόγους χίπηδες οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, κύριε καθηγητά, θα σας συνιστούσα να έρθετε το Μάιο ή Ιούνιο και να δείτε πώς λειτουργεί η σύγχρονη γεωργία στην περιοχή μας στη Βαβαρία. Διότι νομίζω δίνει ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο αηφόρα μπορεί να είναι η γεωργική πολιτική στην Ευρώπη, να διαφυλάσει και το περιβάλλον και να μην έχουμε προβλήματα. η Επιτροπή όπως και κάθε ειδικό, υποτιθέμενος ειδικό, έρχονται να μας κάνουν να μας δώσουν διδαχέ και υπαγορεύσει για το πώς θα πρέπει να καλλιεργούμε τα προϊόντα μας, ενώ εμείς ξέρουμε πολύ καλύτερα από τον καθένα και έχω βαρεθεί να το ακούω αυτό. Το ε, Σαββατοκύριακο μίλησα πάλι με γεωργούς. Έχουμε παραδείγματα όπως ενός νεαρού ε, γεωργού ο οποίος νοικιάζει τα 80 από τα 100 εκτάρια, πρέπει να πληρώνει 800 ευρώ δηλαδή και εάν από αυτά τα 7% πρέπει να ε, μπουν σε αγρανάπαυση θα έχει χάσει 5.600 ευρώ μόνο και μόνο λόγω αυτής της αγρανάπαυσης χωρίς να μπορεί να εκμεταλλευτεί τη γη από τα 80 δηλαδή εκτάρια θα πρέπει να πληρώσει 8.000 επιπλέον ευρώ, συν τα 5.600 που θα είναι χαμένη ευκαιρία καλλιέργειας από τη γη αυτή, δηλαδή κοντά στα 13.500 ευρώ θα πληρώσει για την γη αυτή. Και αυτό που προτείνουν να φύγει το 30%, το 30% για, τα, για την αποθήκευση και το 30% για τη Γενική Διεύθυνση της Γεωργίας και να μας αφήσουν ίσχους να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας και τότε να δει πώς θα μπορέσουμε να εξηγιάνουμε και τον προπολογισμό της ε, Γεωργίας. Εάν λοιπόν ένας νέος Γεωργός μπορεί να δώσει τέτοια, με τέτοια, ε, τέτοια στοιχεία, καταλαβαίνετε πόσο πολύ ανησυχώ για την κατάσταση της Γεωργίας στην Ευρώπη. Ε, Ευχαριστώ, Άλμπερτ, και τώρα Αγνιού. Και κυρία Μάριαν Μαγκίνης μετά. Δεν φαντάζομαι ότι θα μαζέψω χειροκρατήματα όπως ο Άλμπερτ, αλλά και εγώ ήμουν, ε, ε, ασχολήθηκα με αυτό το θέμα το Σαββατοκύριακο. Αν δούμε στην πράξη αυτά τα EFA, το 7% στην δικό μου εκμετάλλευση ήταν 28 εκτάρια περίπου ε, και άλλα 18 που είναι το η επιφάνεια καλλιεργήσιμη θα πρέπει να βγει και κάθε ε, τέτοιο αγρόκτημα θα έχει την ίδια κατάσταση να αντιμετωπίσει. Εν τω μεταξύ πρέπει να θρέψω ένα σωρό κοτόπουλα και αυτό σημαίνει ψηλότερες τιμές ε, για το, τα αυγά στο τελικό καταναλωτή. Ε, αυτό είναι σκανδαλώδε για τον τελικό καταναλωτή. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να βελτιώσουμε τη γη. Ορισμένοι έχουν ε, προβλήματα με το, το, το μαύρο χόρτο, το οποίο όλο ένα και περισσότερο επεκτείνεται και όλο ένα και δυσκολότερο είναι ο έλεγχό του. Ε, ε, να μιλήσω δε για τη βιολογική εκμετάλλευση που έχουν μπει, έχει μπει μάλλον πολύ ψηλά στο βάθρο Πριν από 200 χρόνια αυτό που θεωρούμε πως είναι σήμερα οργανικό και βιολογικό πριν, ε, θεωρεί το ως δηλητήριο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ε, πατάτες. Έχουμε και Εάν όμως ε, εξαρτάται και από τι καιρικέ συνθήκες το τι θα καταφέρεις να κάνεις, υπάρχουν κάποια μηχανήματα τα οποία σκάβουν τόσο πολύ βαθιά ε, που εάν ξαφνικά βρέξει ξεκαταστρέφεται ολόκληρη η καλλιέργεια. Η βιολογική καλλιέργεια δεν είναι το τέλειο και το υπέροχο, δεν πρέπει κανεί να φύγει σκεφτόμενο κάτι τέτοιο. Ε, το έχουμε αλλάξει πολλές φορές ε, το τα προγράμματά μας. Ε, δεν πρόκειται να αλλάξουμε το κλίμα. Εμείς ανταποκρινόμαστε απλώς στις αλλαγές του κλίματος. Μόνο αυτό εξάλλου μπορούμε να κάνουμε. Κάτι, αν πιστεύει κανείς κάτι άλλο, ονειρεύεται. Στη Βρετανία έχουμε επίσης δύο φιλατροπικούς ομίλους ε, τη μία για την προστασία των πτηνών, τον ένα για την προστασία των πτηνών και την άλλη για την ε, προστασία των αγρίων ζώων. Έχουν διαφορετικές ιδέες για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα συμβεί. Το εμπόριο είναι ε, επίσης καλή ιδέα. Οι γεωργοί των Ηνωμένων Βασιλείων το συμπαθούν αυτό γιατί τουλάχιστον μπορούν να αποφασίσουν για κάποια πράγματα ε, πολλοί όμως θα είναι στο πρώτη, στην πρώτη βαθμίδα της, ε, όσον αφορά την, ε, τις υποδιαιρέσεις για τη γη. Βεβαίως ε, θα χτυπηθεί πολύ το Ηνωμένο Βασίλειο. από αυτό το σύστημα αν εφαρμοστεί σε, ολόκληρη τις, σε όλες μάλλον τις γεωργικές περιοχές. Επίσης, περισσότερα προβλήματα θα έχουμε όσον αφορά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Δεν ε, νομίζω πως η Κομισιόν καταλαβαίνει πως αυτό θα χτυπήσει περισσότερο τις, τα μικρότερα, τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις στον Ηνωμένο από ό,τι αλλού. Εάν πρέπει να φυτέψουν ε, κρυθάρι, θα πρέπει ας πούμε να έχουν τρεις φορές ε, συγκομιδή για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Και αν είναι μικροί καλλιεργητές, πάλι δεν θα τα καταφέρουν. Θα πρέπει να υπάρχει η αλλαγή της καλλιέργειας κάθε χρόνο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στα τρία εκτάρια που λέτε. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον δέκα φορές μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Αυτά, Πρόεδρε. Κερδίσατε λίγο έδαφος με μένα. Σας ευχαριστώ, κύριε Άγνιου. Ακόμα και χειροκροτήματα πήρατε. Τώρα η Μάριαν Μαγκίνες και έπειτα η κυρία Κλάς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και όπως και άλλοι θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή Μάθιους για τις προτάσεις του και φαντάζομαι ότι εξ αρχής έχει, ανέφερε κάποια θέματα τα οποία έχω θέξει και εγώ στην Κομισιόν και δεν έχω λάβει απαντήσεις, αν και φαντάζομαι πως θα τις λάβω σε ένα μη έγγραφο, σε ένα non-paper. Ιδιαίτερα όσον αφορά αυτό το πρασίνισμα εξορισμού ε, ορισμένοι συνάδελφοι, πολύ μάλλον συνάδελφοι εδώ, θέλουν ε, να αντιμετωπίζονται ως βιολογικοί καλλιεργητές και άρα το πράσινο συστατικό να καταβάλλεται άμεσα σε αυτούς. Θέλουμε αποσαφήνιση εδώ επιγόντως. Δεν μπορούμε να κινηθούμε προς την υποβολή προτάσεων αν δεν έχουμε προτάσεις από την Κομισιόν για αυτό το θέμα. Και θέλω να συμφωνήσω με τους συναδέλφους ε, με τον ε, Λάινεν για την δημοσιονομική πτυχή, τη σύνδεση με το 30% πρέπει να έχουμε μια πολύ συνεπή πολιτική εικόνα για το τι θέλουμε να κάνουμε. Ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο πιστεύω πως θα πρέπει να κινηθούμε προς την συνειδητοποίηση ότι πρέπει αυτές οι προτάσεις να τροποποιηθούν και να βελτιωθούν. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε καλές πληροφορίες και δεν τις έχουμε ακόμα. Αυτή η παρουσίαση μας βοηθά να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και άρα χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε εδώ. Μια συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά τα σχόλια περί ΠΟΕ. Δεν έχω το νούμερο της διαφάνειας, αλλά το αναφέρατε σε σχέση με το θέμα των προτάσεων πρασινίσματος και διάφορα οριζόντια ζητήματα ας πούμε το θέμα του πράσινου κουτιού. Θα ήθελα να μας πείτε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τις ανησυχίες σας για το συγκεκριμένο ζήτημα και πώς θα μπορούσαμε αυτήν την πτυχή να την ξεπεράσουμε. Εγώ ανέκαθεν έλεγα ότι τα συστατικά, τα πράσινα που προτείνει η Κομισιόν είναι η μικροδιαχείριση των μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων. Εμείς είμαστε κατά αυτούς σε αυτή την Επιτροπή. Θέλουμε οι Γεωργοί να μπορούν να έχουν την ελευθερία να καλλιεργούν, πράγμα το οποίο υποσχεθήκαμε στις τελευταίες μεταρρυθμίσεις. Αυτή η πρόταση είναι αντίθετη προς αυτά όλα. Και γι' αυτό θα θέλαμε λιγότερο να συνδέονται όλα αυτά με τις μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις και ίσως η ιδέα μιας περιφερειοποιημένης προσέγγισης ή ίσως και ακόμα και η εμπορία των EFA θα ήταν κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξει κανείς από τις επιλογές που μας έχετε προτείνει εδώ, γιατί δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για το ποια είναι η καλύτερη πρόταση. Ίσως να μην ε, θέλουν αλλαγές οι συνάδελφοι, αλλά πρέπει να δεχτούμε πώς θα γίνουν αλλαγές και πώς τώρα θα γίνουν αυτές οι αλλαγές από πολιτικής άποψης, από περιβαλλοντικής άποψης και από δημοσιονομικής άποψης αποδεκτές. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μας ανησυχεί όσον αφορά τον αντίκτυπο και ίσως ο καθηγητής Μάθιος θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια παραπάνω για τις συνέπειες. Μιλήσατε για ποσοστά, δεν τα είδαμε στη διαφάνεια. Είπατε ότι θα υπάρξει μικρή, ε, μικρός αντίκτυπος ε, σχετικά για την ε, αρρώσιμη παραγωγή. Τι εννοείτε και είπατε ότι δεν υπάρχει μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Αν στη δεύτερη σας διαφάνεια βλέπουμε ότι το πρασίνισμα είναι αναπόφευκτο δεδομένων των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από το φυσικό περιβάλλον. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η παρουσίαση μας δίνει επιλογές, αλλά δεν μας δίνει την επιλογή να μείνουμε άπρακτοι. Ίσως ο κύριος Μάθιου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα πολιτικό μια πολιτική του ιδιότητα. Οι ακαδημαϊκοί συνήθω δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ήσασταν εσεί στη θέση μα, τι θα κάνατε δεδομένη τη οικονομική σα ανάλυση, ε, του περιβαλλοντικού σας ενδιαφέροντος και των ακαδημαϊκών σας προσόντων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Μάριον, η κυρία Κλά και μετά η Ελίζαμπετ Κόστιντζερ. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Μας παρουσιάσατε μια περιεκτική μελέτη, αλλά είδατε ότι δεν εξαντλούνται οι ερωτήσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε και πολλές άλλες ερωτήσεις, όπως πάντα σε τέτοιους κανονισμούς. Η ε, μετατροπή κατά τρόπο να αξιοποιούνται τα κονδύλια και σε πόσο βαθμό, όπως ρώτησε για κάποιους άλλους βουλευτές, ε, αξίζει με τη μετατροπή αυτή η επιπλέον δαπάνη και το επιπλέον προσωπικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αν ε, ισοδυναμεί με τα αποτελέσματα αυτή η επιπλέον δαπάνη και το κόστος. Επίσης, εκεί όπου ρωτάτε αν αξίζει τον κόπο να γίνει μετατροπή και να περάσουμε σε κανονισμό για να τα εγγράψουμε όλα αυτά. Είπε ο κύριος ε, Ντες ότι δεν αξίζει κάθε ε, επιπλέον μέλος του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην υπόθεση αυτή, γιατί ο κάθε γεωρικός μεταξύ ξέρει πάρα πολύ καλά τι κανόνες και διατάξεις ισχύουν και μπορεί να τις εφαρμόσει μια χαρά. Έτσι λοιπόν έχουμε τόσο πολύ δυσκολέψει, έχει τόσο πολύ επιδεινωθεί η κατάσταση ώστε να μην ε, να θεωρείται ότι κάποιος ε, γεωργός δεν βλέπει αν δουλεύει όχι το σύστημα και αν είναι ικανοποιητικό. Το 7% στο πρασίνισμα. Λέτε με ποια βάση ε, έκτασης θα γίνεται ο υπολογισμός. Στη δική μου την πατρίδα πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν ε, ο υπολογισμός των εκτάσεων. Δηλαδή βγάλαμε χώρο έκταση που καλύπτουν οι ρίζες ενός δέντρου, βγάλαμε το χώρο ή την έκταση που καλύπτει η κήτη ενός ε, μικρού ποταμού, ενός ριακιού και έτσι δώσαμε καθαρή καλλιεργήσιμη έκταση για υπολογισμό. Άλλες χώρε ενδέχεται να μην το έχουν κάνει αυτό. Ε, και άρα θα πρέπει να υπάρξει μια κάποια ισοδύναμη μέτρηση, κάποιο, κάποιο τρόπο, κάποιος τρόπος εξίσωσης αυτών των ε, υπολογισμών. Το 7% ανεκμετάλλευση που αναφέρατε. Στο 7% ανεκμετάλλευση νομίζω ότι πάλι θα οδηγηθούμε σε ε, κατακαιρματισμό της εφαρμογής των μέτρων και απευθύνομαι μεν πάλι προς τους ειδικού. Θα ρωτούσα δεν θα ήταν καλύτερο να υπάρχουν μεγαλύτερες και πιο ενιαίες ε, εκτάσεις, αν θέλουμε να έχουμε σωστά οικολογικά αποτελέσματα, στη τελευταία ανάλυση του Natura 2000 έχουμε κάνει την προσπάθεια ακριβώς για μια δικτύωση των εκτάσεων μέσα στην Ευρώπη. Δεν θα είχε περισσότερο νόημα να προσπαθήσουμε σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο να αναπτύξουμε μια οικολογική ταυτότητα η οποία θα είναι αξιοποιήσιμη και για τον γεωργό και που θα εξασφαλίζει πολύ καλύτερη προστασία από το 7% μιας γεωργικής εκμετάλλευσης που ενδεχομένως θα μπορούσε να ε, ξεχωρίσει ο γεωργός. Και πέραν βέβαια της ε, παραγωγής ε, τροφίμων. Πράγμα που προποθέτει ότι θα έχουμε και επαρκή και καλά τρόφιμα στην Ευρώπη. Άρα ε, άλλη ερώτηση. Υπολογίζονται ήδη οι πράσινες ούτως οικολογικές εκτάσεις που έχουμε ήδη μέσα από το Habitat, μέσα από το Natura 2000, μέσα από τα άλλα συστήματα που ήδη Θα, θα μπορέσετε να κάνετε τη διάκριση. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά λοιπόν, λοιπόν που ε, σας βομβαρδίζω έτσι, αλλά πρέπει να έχουμε σαφείς απαντήσεις για να μπορέσουμε να λάβουμε σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Κόστιγκερ, Πρόεδρε ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστώ ιδιαίτερω και τον καθηγητή Μάθιους για τα πολύ ε, έγκριτα αποτελέσματα που μας προσφέρει από τη μελέτη του. Πρέπει να ομολογήσω ότι είναι δύσκολο να τοποθετηθεί κανείς εδώ σε μια συζήτηση όταν τις απαντήσεις ε, κανονικά θα έπρεπε να τις δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι θα συμφωνήσω και με τους συναδέλφους τις παρατηρήσεις τους και θα επισημάνω ότι θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει και να δώσει σαφείς απαντήσεις ε, ως προς το τι εννοεί σε σχέση με τα μέτρα, ε, ειδικότερα για τις εκτάσεις. Για το δεύτερο πυλώνα, όπου μιλήσατε και όπου Ήδη βλέπουμε κάποιες ε, καλές ευκαιρίες για πρασινίσμα, για μικρά μέτρα, μικρό μέτρα πρασινίσματος. Επειδή μιλάτε για την διαφοροποίηση των μέτρων μέσα στον πρώτο πυλώνα και μέσα στον δεύτερο και λέτε παντότε ότι θα πρέπει να μένουν χωριστά τα μέτρα του ενός πυλώνα από εκείνα του άλλου. Εδώ έχουμε να κάνουμε μέτρα τα οποία σε ένα βαθμό έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη-μέλη και αφορούν το πρασίνισμα και μέσα στον, πράσινο, στον πρώτο πυλώνα. Ερωτώ λοιπόν σε σχέση με το, screen, με το πρασίνισμα το οποίο πρέπει να περάσει στον, στον δεύτερο πυλώνα, πώς βλέπετε την εφαρμογή ε, και τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων αυτών. Όλα αυτά το, τα οποία ονομάζονται πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του δεύτερου. Θα είναι ακόμη εκούσια. Στην ε, Αυστρία έχουμε περίπου 90% των γεωργών που δέχθηκαν να υπαχθούν στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Άρα βλέπουμε πόσο μεγάλη υποδοχή είχε αυτό το μέτρο, αυτή η δυνατότητα. Αλλά θα ήθελα εδώ να ε, επισημάνω εκ προημίου ότι χρειάζεται διαφορετική και θα χρειαστεί διαφορετική πλαισίωση εφόσον εισαχθούν διαφορετικά μέτρα πέραν δηλαδή του, των αγροπεριβαλλοντικών. Επίσης το 10% της μεταφοράς από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Εκμεταλλεύσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για τα αγροπεριβαλλοντικά. Πώς θα σας φαινόταν εάν βγαίνανε αυτομάτως από το πρασίνισμα. Ευχαριστώ, Πατράου Ναβέσου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον καθηγητή Μάθιου που μας βοήθησε εδώ για να σκεφτούμε το θέμα του πρασινίσματος. Ήδη υπόθηκε ότι χρειαζόμαστε κάποιες ακόμα απαντήσεις από πλευράς της Κομισιόν, ώστε να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να λάβουμε τις καλύτερες πολιτικές αποφάσεις. Από αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής υπάρχουν τρία, από όσα μάλλον μέχρι στιγμής, εγώ θα ήθελα να τονίσω τρία πράγματα. Το πρώτο και είναι το θέμα το περιβαλλοντικό για το οποίο μιλάμε. Πρόσφατα άκουσα έναν πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λέει ότι η μεταρρύθμιση έχει στόχο να τοποθετηθεί το περιβάλλον στο επίκεντρο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εγώ συμφωνώ απόλυτα πως τα μέτρα, τα περιβαλλοντικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και ότι πρέπει να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με αυτά. Όμως εγώ ρωτώ, μέχρι ποιο βαθμό αυτός ο εστιασμός ο κρέος στα περιβαλλοντικά θέματα μπορεί να μας οδηγήσει στο να χάσουμε από την, οπτική μας ε, γωνία ε, αυτό που είναι το βασικό στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής, δηλαδή η παραγωγή τροφίμων. Έχουμε πολύ σημαντικό θέμα, την επάρκεια. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες ε, τροφίμων μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό όπλο και γι' αυτό λέω προσοχή. Προσοχή μην ξεχάσουμε αυτό που πραγματικά βρίσκεται στην βάση της γεωργικής ε, πολιτικής, δηλαδή η παραγωγή τροφίμων και κυρίως η επάρκεια σε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα αφορά την ισότητα. Την ισότητα που είναι η βάση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και που ε, αναφέρεται με ιδιαίτερο τρόπο όταν μιλάμε για πρασίνισμα. Θα έχουμε ένα ενιαίο πρότυπο για τις 27 χώρες μέλη. Αν ε, γίνει κάτι τέτοιο θα ήταν ε, πολύ καλύτερα προσαρμοσμένο για κάποιους και πολύ λιγότερο προσαρμοσμένο για κάποιους άλλους. Και άρα λοιπόν η ισότητα παραβιάζεται άμεσα. Τι γίνεται με την άρδευση, για παράδειγμα, που είναι πολύ ουσιαστική για όλες τις ε, νότιες χώρες και να μην ξεχνάμε πως αυτή τη στιγμή διανύουμε μια ε, εξαιρετικά έντονη ε, λειψιδρία. Εάν δεν γίνεται άρδευση, με κάποιο τεχνολογικό και περιβαλλοντικό τρόπο δεν γίνεται να έχουν καλλιέργεια οι νότιες ε, γεωργία, συγγνώμη, οι νότιες χώρες. Ε, οπότε πού είναι η ισότητα. Και έπειτα Υπάρχουν και κάποιες περιοχές οι οποίες εξαρτώνται από τη γεωργία για να μπορέσουν να διατηρήσουν την πυκνότητα του πληθυσμού τους. Θα έχουμε συγκεκριμένα μέτρα, ειδικά μέτρα για την ιδιαιτερότητα αυτών των λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Κάτι τέτοιο θα είναι πολύ σημαντικό για να διατηρηθεί η ισότητα. Και έπειτα, αν μιλήσουμε πάλι για ισότητα, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ισότητα, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για δίκαιο πρασίνισμα, αν η ίδια η ανακατανομή δεν είναι δίκαιο Εάν ξέρουμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν χώρες ε, τη σήμερον ημέρα όπου, το, όπου η Πορτογαλία λαμβάνει, ας πούμε, ε, πολύ λιγότερα από χώρες που παίρνουν 400 ευρώ ανά εκτάριο. Πώς θα γίνει το πρασίνισμα με αυτό το 30% είναι ίδιο το 30% σε όλα τα κράτη-μέλη ή ανάλογα με την απόδοση του κάθους, κάθε κράτους μέλους γιατί ακριβώς η ίδια η ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων είναι διαφορετική. Γι' αυτό και νομίζω ότι το θέμα της ισότητας είναι ανοιχτό. Τελευταία μου παρατήρηση με όλα αυτά τα μέτρα πρασινίσματος στον πρώτο πυλώνα, όπως υπόθηκε και από τον καθηγητή Μάθιου, ορισμένα μέτρα είναι πολύ κοντά στη δεύτερο πυλώνα, ενδεχόμενη επικάλυψη, ενδεχόμενη ε, διπλασιασμός τελικά. Μήπως φτάσουμε στο 1 τρίτο μόνο, δηλαδή στην απλοποίηση, που είναι σημαντική είναι σημαντική όχι μόνο για τους ε, γεωργούς αλλά και για την ε, δημόσια αποδοχή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα ο Ζωζέ Μποβέ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καλά την πραγματική κατάσταση όσον αφορά την υποβάθμιση του γεωργικού περιβάλλοντος. Και εδώ δεν μιλάω για τον κήπο που μπορεί να είναι η Αυστρία ή η Βαβαρία. Αυτές είναι χώρες καλά ισορροπημένες, δεν μιλάω για αυτό. Αλλά για πηγαίνετε σε κάποιες παιδιάδες όπου καλλιεργούνται δημητριακά στη Γαλλία για παράδειγμα ή στη Ρουμανία ή σε άλλα γερμανικά κρατήδια στο βορρά της Γερμανίας η κατάσταση είναι τραγική εξαιτίας των νητρικών, εξαιτίας ε, ε, των ε, φρεατίων, των υπόγειων υδάτων κλπ. Είναι απειλές για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε στα σοβαρά αυτό το θέμα, το θέμα της εκπεριτροπής καλλιέργειας, ώστε να βελτιωθεί αισθητά η κατάσταση. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε ανάλυση αντικτύπου για αυτά τα μέτρα. Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια πραγματική ανάλυση αντικτύπου από την εκπεριτροπή καλλιέργεια. Δεύτερο, μπορεί να μιλάμε για τη γραφειοκρατία, αλλά και εδώ ας σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν χώρες όπου ε, η κοινή γεωργική πολιτική αναλύεται και υπάρχουν μέσα αποτελέσματα. Άρα έχει γίνει επαλήθευση σε ορισμένες χώρες μέλη όσον αφορά την εκπεριτροπής ε, καλλιέργεια. Και θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο μέτρο να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε αυτονομία όσον αφορά τις ζωικές πρωταΐνες. Αν συμπεριλάβουμε ως κύριο στόχο της εκπεριτροπής καλλιέργεια την επίτευξη της ε, αυτάρκειάς μας, σε φυτικές πρωτεΐνες, σε πρωτεΐνες, τότε αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Έπειτα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Εδώ και καιρό ακούω διάφορα για αυτό το 30% και το πρασίνισμα. Και πολλές χώρες μέλη αντιτίθενται. το να θέλουμε να έχουμε επιλογές αλλά καρτ και το κάθε κράτος μέλος να έρχεται και να παίρνει το ένα ή το άλλο, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να σαμποτάρουμε την πρόταση. Γι' αυτό να είμαστε αυστηροί και απόλυτοι και να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει κοινή θέση, συλλογική και να βγούμε από τη λογική αυτή που λέει ότι κάθε χώρα μέλος θα κάνει αυτό που θέλει, δηλαδή θα λέει ε, να αλλάξουν οι άλλοι, εγώ δεν θα αλλάξω και ας έχουμε καταστροφή μεθαύριο, δεν πειράζει. Τζανκάρλο ε, Σκοτά. Ναι, με συγχωρείτε. Εγώ εν μέρει συμμερίζομαι τα όσα είπε αρχικά ο Μποβέ. Ξεκίνησε πολύ καλά λέγοντας ότι κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της και ότι τα κράτη-μέλη το καθένα έχει δεσμευθεί λιγότερο ή περισσότερο για το ποια είναι η ε, γεωργική επιφάνεια. Αλλά το να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο σύστημα με βάση για, το ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή επικρότητα είναι λάθος. Ίσως θα πρέπει να επιβάλλουμε κανόνες στα κρατημέλη ώστε να ε, σέβονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους τι θα είναι αυτό το πρασίνισμα που θα εφαρμοστεί στις γεωργικές περιοχές. Και δεν καταλαβαίνω τι, το πώς θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα συντονίσουμε σε κάποιες περιοχές, σε ορισμένε ζώνε όπου έχουμε εντατική καλλιέργεια α πούμε, ενώ αλλού έχουμε ε, κήπου ωραιότατου. ωραία. Ε, μπορούμε εκεί να παρεύουμε και πολύ πιο έντονα, αλλά σε ένα σωρό σημεία, σε πολλές ζώνες υπάρχουν εγκαταλελειμμένες περιοχές. Αυτό το πρασίνισμα δεν θα πρέπει να γίνει, όπως είπε πριν η Κράς, κάθε ε, μέρος το οποίο χρησιμοποιείται ε, και μετά θα το παρατήσουν και θα εγκαταλειφθεί ακριβώς και μόνο για να πάρουν το greening αυτό που λέμε. Πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί αυτό το greening, εντάξει, αλλά μετά να αξιολογήσουμε την ε, πτυχή, τη χωροταξική του κάθε κράτους για να μπορέσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εντοπίσουμε τους στόχους. Γιατί όλοι, όλους, όλοι θέλουν να συντηρήσουν το περιβάλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ε, φτιάξουμε ένα ενιαίο πράγμα ενώ υπάρχουν τόσο πολλές ιδιαιτερότητες. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Καθηγητά Άλαν Μάθιο, πιστεύω πως ε, ακούσατε μια πολύ μεγάλη ε, ένα μεγάλο φάσμα ερωτημάτων ε, και απόψεων και εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω υπό το φως ε, της εξαίρετης αυτής παρουσίαση την οποία εκτίμησα όλος ιδιαίτερος λαμβάνοντας υπόψη ότι καθένας δεν είναι αντίθετος ε, στη σχέση με Ε, σε σχέση με την οικολογική, τον οικολογικό χαρακτήρα. Όμως ανησυχούμε για το αν όλοι οι Ευρωπαίοι Γεωργοί θα καταφέρουν να εφαρμόσουν ε, τους κανόνες του greening που προβλέπει η Κομισιόν. Στην πιο αισιόδοξη υπόθεση, αν θα είναι το 90% των Ευρωπαίων Γεωργών, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι πάνω από 4 δις ευρώ θα επανέλθουν στην ευρώ, στην, ε, στις Βρυξέλλες. Η Υπό το φως λοιπόν όλων αυτών των προβληματισμών και του θέματος της επιστημιστικής ασφάλειας που σίγουρα είναι θεμητό πέρα από το περιβαλλοντικό, την περιβαλλοντική πτυχή, ποιο είναι ο τρόπος κατά τη γνώμη σας που θα μπορούσαμε εμείς ως Κοινοβούλιο να προτείνουμε ώστε να επιτύχουμε το 100% του πρασινίσματος στους Ευρωπαίους Γεωργούς. Σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να μείνετε στα 10-12 λεπτά στην απάντησή σας. Ευχαριστώ. Well, <coughs> can I... Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά εγώ δεν εκπροσωπώ εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές από τις ερωτήσεις σας απευθύνονταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά επιτρέψτε μου να σχολιάσω παρόλα αυτά κάποια πράγματα. Θα παίρνει φυσικά πάρα πολύ χρόνο να προσπαθούσα να απαντήσω χωριστά στην κάθε ερώτηση που ακούσαμε. Ορισμένες έτσι κι αλλιώ συμπεριλαμβάνονται στο σημείο μου. Απλώ εγώ δεν είχα καιρό να σας τα παρουσιάσω όλα. Όποιο ενδιαφέρεται και έχει χρόνο πάντως μπορεί να ε, διαβάσει το σημείωμά μου. Θα επικεντρωθώ σε τρία σημεία όμως, τα οποία ακούστηκαν ξανά και ξανά. Το ένα έχει να κάνει με τον πυλώνα 2, το δεύτερο είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, συνδέονται εξάλλου, και το τρίτο ήταν ο ορισμός του πρασινίσματος και το θέμα των βιολογικών καλλιεργιών. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω κυρίως σε αυτά τα τρία και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις που ακούστηκαν. Ο κύριος ε, Λάιον είπε, είπε ότι αν ξεκινούσαμε από την αρχή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξεκινούσαμε με την πρόταση που έχουμε τώρα μπροστά μας. Μα η κοινή γεωργική πολιτική έχει πράγματι μια ιστορία, 50 χρόνια πίσω της. Συνεπώς αυτό σίγουρα περιορίζει κάπως την κατεύθυνση που παίρνει η πολιτική μας. Είναι χρήσιμο όμως να σκεφτούμε ότι 30% των εθνικών οροφών είναι κάτω από 13 εκατομμύρια το χρόνο και ότι αν είχαμε 13 δις το χρόνο για να βοηθήσουμε τους αγρότες να καλλιεργούν ε, πιο περιβαλλοντικά, θα έπρεπε να δούμε τι θα είμαστε διατεθειμένοι να ξοδέψουμε. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δηλαδή, τι κάνουμε για να τροποποιήσουμε τον κανονισμό που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, σεβόμενοι κάποιες αρχές που υπάρχουν ήδη και προκειμένου να υπάρξουν απαντήσεις στις προτάσεις της Επιτροπής, θα ήταν χρήσιμο να δούμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Απόψη μου είναι ότι πολλά μπορεί να πει κανεί για τον πυλώνα 2. Τα αναφέρατε κι εσείς. Είναι σε θελοντική βάση και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αν θέλουμε να έχουμε ε, περισσότερη περιβαλλοντική διάσταση στην γεωργία μας, ε, θα έπρεπε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τη γη. Το ότι νιώθουν οι αγρότες ότι τους επιβάλλουμε ε, τις διατάξεις αυτές, ότι τους έρχονται απ' έξω και νιώθουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αυτό όντως είναι αρνητικό. Αντίθετα, θα έπρεπε να στερνίζονται τις ρυθμίσεις αυτές και να νιώθουν ότι όντως ε, είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν στο πρασίνισμα. Γι' αυτό και πρέπει να δουλέψουμε με τους αγρότες. Πρόκειται για μια πολυετή ρύθμιση, οπότε περιβαλλοντικά αυτό έχει πλεονεκτήματα. Επίσης είναι στοχευμένα μέτρα, γιατί μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα ενός περίπλοκου μενού, όπως είπαμε, και όλα αυτά μπορεί κανείς να τα διαχειριστεί στα πλαίσια του πυλώνα 2. Αν βέβαια αποφασίσετε να συνεχίσετε το πρασίνισμα στον πυλώνα 1, τότε περιορίζετε τις επιλογές σας. Οι λόγοι πάντως που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι οι υπερβαλλοντικοί κανόνες πρέπει να είναι απλοί, γενικευμένοι και αιτήσιοι. Οπότε αυτόματα περιορίζουμε τον οριζοντά μας πάρα πολύ. Πάντως, ενδιαφέρον είναι να δούμε και το θέμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του ΠΟΕ. Κάποιοι ομιλητές είπαν ναι, αλλά αν έχουμε διαφοροποίηση στη σοδιά, δεν θα έπρεπε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο και να ξέρουμε για ποιες σοδιές μιλάμε. Μα στα μέτρα τύπου πυλώνα 1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα πρόκειται για μια ενίσχυση εισοδήματος στο Green Box Και αν συνδέσετε την πληρωμή από τον πυλώνα 1 σε οτιδήποτε το οποίο να φαίνεται να είναι απέτηση για μείωση της οδειάς, τότε δεν ε, μπορείς να ισχυριστείς ότι πρόκειται για πληρωμή green box. Βέβαια κάποιοι ρώτησαν, είπαν αν υπάρξει εξαίρεση για τις βιολογικές καλλιέργειες, μήπως αυτό τελικά απειλεί το καθεστώς ε, του πράσινου κουτιού και τις πληρωμές πρασινίσματος από εκεί. Αυτό το εξηγώ στο σημείωμα, αλλά κυρίως κοιτάω κατά πόσο η διαφοροποίηση στις σοδιές απειλεί το καθεστώς ε, αυτό green box στις πληρωμές. Και εγώ βέβαια βλέπω κάπως πιο ουδέτερα τα πράγματα από ότι ο καθηγητής ε, Σλίμπαρκ. Αυτά τα πράγματα είναι όντως πάρα πολύ δύσκολα για να τα προβάλλει κανείς στο χρόνο. Έχω συμμετάσχει στον ΠΟΕ μερικές φορές, παρόλα αυτά δύσκολα μπορεί κανείς να προβλέψει. Πάντως, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε στα πλαίσια της διαφοροποίησης της στοδιάς ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή και μιλάω τώρα για ότι είναι συμβατό με τον ΠΟΕ, έτσι και όχι για άλλα επιχειρήματα. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή είναι να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραγωγή. Δηλαδή δεν λέει ότι πρέπει να έχεις αυτή την καλλιέργεια την άλλη, αλλά λέει ότι αν έχεις μία καλλιέργεια τότε εμεί απαιτούμε να έχεις διαφοροποίηση στο μοντέλο καλλιέργειας της γης σου. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραγωγή δηλαδή. Δεν υπάρχει απέτηση για συγκεκριμένη παραγωγή του ενός ή του άλλου προϊόντος. Και με τα βιολογικά προϊόντα και εδώ έχουμε να κάνουμε με τη διαδικασία παραγωγής. Και ο ΠΟΕ, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει να αναμειχθεί σε αυτό. Εκτός αν το είδος της καλλιέργειας έχει να κάνει με το είδος παραγωγής του, με τον τρόπο με τον οποίο παράγεται. Εμένα όντως με ανισχούν πάντως τα μέτρα του ΠΟΕ που ισχύουν ήδη και η σχέση με τις προδιαγραφές ΓΑΕΚ. E Και έχει τόσο οτιδήποτε νέο προσθέτει πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκτός βέβαια από τα μόνιμα βοσκοτόπια. Γιατί εδώ ο κίνδυνος μπορεί να είναι να ευνοείται ε, το ένα ή το άλλο είδος γης. Είναι ενδιαφέρον πάντως το ότι αν συνεχίσουμε και εξετάσουμε τα θέματα αυτά βάσει του, πυλένα, του πυλώνα 2 για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, τότε αποφεύγουμε πλήρως το θέμα του ΠΟΕ. Γιατί άπαξ και καλύπτει στα γενικά κριτήρια για αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα που αποζωμιώνεται ο αγρότης για τα έξοδά του, πρόκειται για καθαρά περιβαλλοντικά προγράμματα, τότε τα ειδικά μέτρα για όσπρια ή οτιδήποτε άλλο δεν έχουν νόημα. Στην περίπτωση του πυλώνα 2 δεν έχει νόημα αυτό, οπότε υπάρχουν άλλα πλεονεκτήματα στον πυλώνα 2 εκτός από αυτά τα οποία αναφέραμε ήδη. Κάποιοι ομιλητές, και καταλαβαίνω γιατί, αναφέρθηκαν στη γραφειοκρατία και στην διοικητική περιπλοκότητα. Άποψή μου είναι ότι εάν θέλουμε να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε κίνητρα και κανονισμούς στην γεωργική μας πολιτική προκειμένου να πείσουμε τους αγρότες και όσους διαχειρίζονται τη γη να πάνε προς μία πιο αηφόρο κατεύθυνση, πιο περιβαλλοντική, ε, σίγουρα αυτό θα απαιτήσει επιπλέον γραφειοκρατικό κόστος. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό. Και έτσι ερχόμαστε πίσω στο πιο γενικό θέμα που λέει «Α, δεν θέλουμε καμία σχέση με το πρασίνισμα». Τότε ο προϋπολογισμός για τις άμεσες πληρωμές διακινδυνεύεται. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να καταδικάσουμε την πρόταση απλώς και μόνο επειδή απαιτεί μία επιπλέον διοικητική προσπάθεια, γι' αυτό και μόνο. Όχι, πρέπει να δούμε πόση παραπάνω γραφειοκρατική προσπάθεια, διοικητική μάλλον προσπάθεια χρειάζεται. Τι βλέπουμε εμείς ως ε, όφελος από αυτά τα μέτρα, όφελος για το περιβάλλον, παρά το διοικητικό άχθος. Νομίζω ότι τα ειδικά μέτρα εξαιτία της φύση τους ακριβώς, γενικευμένα μέτρα, προσφέρουν περιορισμένα περιβαλλοντικά ωφέλη. Είπαμε που είναι τα μεγαλύτερα ωφέλη. Το θέμα του σε τι βαθμό έχουμε τέτοια ωφέλη και σε τι βαθμό μπορείς να επιτρέψεις επιπλέον ελαστικότητα στα κράτη-μέλη χωρίς να καταλήξεις ένα σύστημα à la carte. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην μπορεί κανείς να αποφύγει τις υποχρεώσεις του. Πώς δηλαδή καταλήγει σε ισοδύναμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη η οποία θα πρέπει να αποφασίσει. Δηλαδή έρχονται τα κράτη-μέλη με τα προγράμματά τους, τα οποία αξιολογούνται ως ισοδύναμα τουλάχιστον της βασικής γραμμής που περιλαμβάνεται στη ρύθμιση. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές διαστάσεις περιβαλλοντικής ε, προσπάθειας και περιβαλλοντικού αποτελέσματος που θέλουμε να ενθαρρύνουμε. Συνεπώς, Κύριε Μαγκίνες, τι θέση σας διαθετούσα κι εγώ. Και αυτό είναι το καλό όταν κανείς είναι ακαδημαϊκός. Είναι ότι μπορεί να δει τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Σαν κάποιος απ' έξω θα λέγα ότι αυτό το οποίο εκπλήσει λίγο είναι ο στόχος και η μετακίνηση από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2. Πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν την προσπάθεια που γίνεται στον πυλώνα 1 και στον πυλώνα 2. Πάντως, αν δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Αν υπάρξει επιπλέον προϋπολογισμός που θα περάσει από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 και εδώ δεν υποτιμάω τις δυσκολίες που υπάρχουν, όπως το θέμα της συγχρηματοδότησης που αναφέρθηκε ήδη. Τα κράτη-μέλη εθελοντικά, άραγε θα έπρεπε να μετακινηθούν από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα επιτραπεί κάποια ελαστικότητα. Επιπλέον με το 10% την ε, εθελοντική διαφοροποίηση. Υπάρχουν ε, τρόποι πάντως για να αυξηθεί ο προπολογισμό του πυλώνα 1. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το επιθυμητό και το επιδιωκόμενο. Πάντω δέχομαι και το επιχείρημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής που λέει τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του πυλώνα 2 σε μερικές χώρες πράγματι υπάρχει παντού κάλυψη, σε ολόκληρη τη χώρα, όπως στην Αυστρία. Αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, που και σωστά ίσως είναι περήφανη για τα αγροπεριβαλλοντικά της προγράμματα, λιγότερο από το 50% της γης περιλαμβάνονται σε τέτοια προγράμματα. Το άλλο 50% όχι. Και ακριβώς αυτό το 50% είναι που στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που δεν καλύπτεται από αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα. Συζητάμε λοιπόν για το πώς θα αυξήσουμε τον ε, πύχη παντού Πέρα λοιπόν το ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα με τον πυλώνα 2, καλό θα ήταν να δούμε μήπως μπορούμε τη βασική γραμμή να την ανεβάσουμε, τον πύχη να τον ανεβάσουμε. Ξέροντας ότι οι προδιογραφές ΓΚΑΙΚ e προσφέρουν κάποια ελαστικότητα στα κράτη-μέλη. Δεν είναι άκαμπτοι κανόνες, δεν είναι ομοιόμορφοι. Υπήρξαν επικρίσεις κατά το παρελθόν, αλλά για μένα, έχοντας εξετάσει τις διάφορες προτάσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει μία πρόταση η οποία να τα πετυχαίνει όλα και δικαιοσύνη και οικουμενικότητα και αποτελεσματικότητα και χαμηλό διοικητικό κόστος και καλά περιβαλλοντικά ωφέλη. Μπορεί λοιπόν να αξίζει κάποιο παζάρεμα. Να αυξηθούν οι προδιαγραφές, αλλά από την άλλη μεριά τα κράτη-μέλη να μπορούν να καθορίσουν πώς θα εφαρμόζουν τις προδιαγραφές αυτές στο καθένα στον τόπο του και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του. Ευχαριστούμε καθηγητά Μάθιους. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Και τώρα σύντομα πρέπει να καλύψουμε χρόνο. Να πάμε στο σημείο 5 της σημερινής ημερησίας διάταξης. Να αποχαιρετήσουμε τον καθηγητή. 5 λοιπόν, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων. Όχι, πήδηξε ένα. Τέσσερα πρώτα. Κοινή οργάνωση αγορών των χειρουργικών προϊόντων. Η κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ. Δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ μετά από την πρώτη συζήτηση που έγινε στις 23 Ιανουαρίου που μας πέρασε και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να θυμίσω σε όλους ότι θα έχουμε δύο ειδικά εργαστήρια σε σχέση με το κόα 27 Μαρτίου το απόγευμα. Ε, θα έχουμε μια παρουσίαση για τους μηχανισμούς του ΚΟΑ και τα μέσα διαχείρισης του κινδύνου. Και έπειτα θα έχουμε ένα δεύτερο εργαστήρι στις 24 Απριλίου το απόγευμα μια παρουσίαση του πλαισίου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συγκεκριμένων κανόνων για την ε, τροφιδιατροφική αλυσίδα μέσα στο πλαίσιο της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής. Μπαίνουμε στο πυρήνα του θέματος δηλαδή. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Μισελ Νταντά και μετά βεβαίως θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. η συζήτηση προηγούμενη σκέφτηκα ότι σας οδήγησε τόσο βαθιές σκέψεις που με ξεχάσατε. Αλλά για την οργάνωση θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι η τρίτη φορά που περιστέλλεται ο χρόνος που αφιερώνουμε στις, ε, στις ΚΟΑ και μάλιστα κατά μισή ώρα αυτή τη φορά. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η δέσμη μέτρων που έχουμε μπροστά μας ε, απαρτίζεται κατά με από τέσσερις ε, κατηγορίες. Η πρώτη, την οποία θα μπορούσα και να διαγράψω στικά γιατί βλέπω ότι συμφωνούμε όλοι, έχει να κάνει με τα τομεακά ζητήματα, δηλαδή ε, θέματα ίνου, σακχάριος και γάλακτος. Για, το γάλα και τον, για τη σάκχαρη και τον ε, ίνο έχουμε λίγο πολύ συμφωνήσει και από τις συζητήσει που είχα με εκπροσώπους των δύο τομέων όπου επεσήμανα ότι δεν ε, βλέπω εύκολο να προβλεφθεί πρόταση για παράταση των προθεσμιών ανεφετέρου. Άρα θα χρειαστείτε μια σταδιακή ε, κατάργηση για τη ζάχαρη ή μια ε, διαφορετική διαδικασία όμοια σε όλα τα κράτη, ενωποιημένη δηλαδή, ε, για τον Νίνο και βέβαια τις σχετικές προτάσεις θα τις ε, διατυπώσω εφόσον έχω ακούσει και όλες τις πλευρές. Ε, δεύτερο κεφάλαιο, τα μέτρα για αντιμετώπιση κρίσεων, κανόνες ανταγωνισμού, σχέση μεταξύ παραγωγών. Στα μέτρα ανταγωνισμού είπατε και εσείς πρόεδρε ότι 24 Απριλίου, γιατί πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατηγορία, θα έχουμε συζήτηση με τους ειδικού και το θέμα αυτό θα το άφηνα κατά μέρος για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο. Θα ήθελα να αναλογιστούμε από κοινού και να ακούσουμε τις διαφορετικές απόψεις. Πιο πολύ στα μέτρα ε, αντιμετώπισης κρίσεων και της οργανώσεις των παραγωγών τα μέτρα αντιμετώπιση κρίσεων στο κείμενο που μα προτείνονται δεν αποτελούν τίποτα καινούριο. Δηλαδή, επαναλαμβάνονται προτάσει που ήδη υπήρχαν, που απλώ μερικέ φορέ ε, λησμονήθηκε η επικαιροποίησή του ε, ή ο εξυγχρονισμό του. Σε πάση περιπτώσει, θα το προσπαθήσουμε εμεί αυτό. Αλλά εισάγεται η έννοια αυτού του ε, δικτύου ασφαλεία μια ιδέα μια έννοια η οποία έχοντας ακούσει και τους άλλους διαπιστώνω ότι μπορεί να ε, σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθέναν. Και θα ήταν καλό να ε, συζητήσουμε πώς βλέπουμε ο καθένας μας αυτή την ε, έννοια δικτύου ασφαλείας. Δηλαδή τι εννοούμε όταν ακούμε δίκτυα ασφαλείας. Ένα από τα υποτείνοντα στοιχεία αυτή τη μεταρρύθμιση είναι η απουσία τη της κρατική παρέμβαση, η λειτουργία δηλαδή των αγορών και κυρίω μέσα ε, από, την αλυσίδα των προϊόντων. Και το θέμα είναι θέλουμε πραγματικά να προβάλλουμε αυτήν την ε, επιλογή, θέλουμε να αφήσουμε δηλαδή, στην αλυσίδα του προϊόντος να αφήσουμε να επαφίεται η διαχείριση του τομέα και αν ναι, δεν θα πρέπει να προσδιορίσουμε μέσα και δυνατότητες γιατί δεν αρκεί βέβαια να διατυπώνουμε μια βούληση και μετά να παραμένουμε στις παλές πρακτικές και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα ούτε οι οργανώσεις παραγωγών ούτε η, η αλυσίδα της παραγωγής. Ε, το ίδιο ισχύει και για, τους, για τις ενώσεις των παραγωγών. Δεν προσπαθούμε βεβαίως να θεσπίσουμε νέες ή να εφεύρουμε νέες δομές παραπέμπουμε στο εθνικό δίκαιο. Κάθε κράτος ορίζει ως ένος παραγωγών αυτό που θεωρεί σκοπιμότερο να ορίσει ως ένας παραγωγών. Συνήθως εννοούνται οι συνεταιρισμοί, αλλά ακόμα και με την έννοια του συνεταιρισμού κάθε κράτος μπορεί να έχει διαφορετική αντίληψη. Και γι' αυτό καλό θα ήταν η Επιτροπή μας μέσα από μια ε, έκθεση πρωτοβουλία, να αναλογιστεί τι εννοεί με την έννοια του συνεταιρισμού της ένωσης των παραγωγών, τι σημαίνει σε κάθε χώρα αυτή η Ένωση Παραγωγών Εσωτερετηρισμός. Και πάλι τι τίθε το ζήτημα τι, κάνουμε, ε, τι, τι δυνατότητες δίνουμε στις ενός παραγωγών, όπως είχαμε κάνει με το γάλα, τη δυνατότητα για διαπραγμάτευση συμβάσεων, τιμών ενδεχομένω ε, που θα πρέπει να επεκταθεί ερωτηματικό σε όλες τις παραγωγές, σε κάθε τομέα παραγωγή και μπορεί η Ένωση Παραγωγών να ρυθμίσει ε, μια αναγορά και τις ε, ικανότητες παραγωγής, του δυναμικό παραγωγής. Επίσης, σε ποιο βαθμό η γεωργική παραγωγή μπορεί να έχει την πρόσβαση αυτά τα ε, σημαντικά δημοσιονομικά μέσα που είχαν θεωρηθεί ως πανάκια μεν που όμως αποδεικνύεται ύστερα από προσεκτική θεώρηση ως ένα δαπανερό εργαλείο και μάλιστα προσβάσιμο μόνο σε ορισμένους παραγωγούς και όχι σε όλους. Και άρα θα πρέπει να ρωτηθούμε τι μέσα θέλουμε να προσφέρουμε στο Γεωργό ώστε να μπορεί να προσφεύγει, να αξιοποιεί αυτά τα νέα μέσα, τα δημοσιονομικά μέσα. Αυτά είναι η βάση της συζήτηση, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Μισελ. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση και δίνω το λόγο στην κυρία Γκαρσία Περέση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σημερίζομαι τις περισσότερες παρατηρήσεις που έκανε ο εισηγητής. Θέλω όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα, τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να τα δούμε πιο συγκεκριμένα και να επιμείνουμε σε αυτά και να δούμε μήπως η Κομισιόν μπορεί να μας βοηθήσει εξηγώντα μας τι ακριβώς συμβαίνει. Για τα μέτρα παρέμβασης, για παράδειγμα, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πραγματικό δίκτυο ασφάλειας που να έχει να κάνει με έκτακτα μέτρα σε περίπτωση ιδιαίτερων κρίσεων. Μην ξεχνάμε ότι σε κάθε τομέα μπορεί να υπάρξει τέτοια κρίση που να δικαιολογεί έκτακτα μέτρα και δεν μπορούμε να βγάλουμε καμία παρέμβαση από εδώ. Ιδιαίτερα μάλιστα να διευρύνουμε και τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα συμπεριλαμβάνοντας περισσότερα προϊόντα με στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον κάθε τομέα. Τώρα τα μέτρα από την άλλη μεριά πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή αυτόματα. Ιδιαίτερα πρέπει να δούμε τις τιμές που έχουν να κάνουν με το ελαιόλαδο και με τα οποροκυπευτικά. Σίγουρα σε περίπτωση που έχουμε κρίση πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά ποσά και μηχανισμοί που επιτρέπουν αποτελεσματικά και γρήγορα να αντιμετωπίζονται διακοιμάνσεις στην αγορά. Δεν ξέρω τώρα έτσι όπως ε, μιλάει, έτσι όπως το διατυπώνει μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα ταμείο κρίσης θα μπορούσε ε, γρήγορα να ανταποκριθεί σε περίπτωση προβλήματος. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή μας. Το ένα είναι ταμείο κρίσης, το άλλο είναι αποθεματικό κρίσης. Δεν ξέρω, πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω. Θα μπορούσε και το ταμείο να αντιδράσει τόσο γρήγορα. Για τέκτακτα μέτρα τώρα σε περίπτωση ε, προβλημάτων στην αγορά, έχουν ε, μπει στο βλάκι, αλλά πρέπει αυτόματα να μπαίνουν σε εφαρμογή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Τώρα όσον αφορά ε, τις προδιαγραφές εμπορίας, ξέρετε ότι εδώ πρόκειται για διάφορα ε, στοιχεία και ότι η Επιτροπή μας έχει ήδη οθετήσει μέτρα τον Ιούλιο με το πακέτο ποιότητας. Δεν καταφέραμε όμως να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και ακόμα δεν έχουν εντολή για να ξεκινήσει ο διάλογος. Συνεπώς η συμφωνία που πετύχαμε με τους συζητητές των άλλων πολιτικών ε, ομάδων έχει σαν αποτέλεσμα το πακέτο στο οποίο θα καταλήξουμε αυτόματα να συμπεριληφθεί στην έκθεση του κυρίου Νταντάν με τις δικές μας ε, τροπολογίες. Η βελτίωση τώρα της λειτουργίας ε, των διαδικασιών εμπορίας είναι κάτι που πρέπει να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το πακέτο με τα γαλακτοκομικά και το ελαιόλαδο. Όλοι οι τομείς πρέπει να, για όλους τους τομείς πρέπει να αναγνωρίζουμε τις επαγγελματικέ ε, οργανώσεις του κάθε κλάδου και να λάβουμε υπόψη μας το θέμα της συγκέντρωσης της προσφοράς, την εμπορία και την παραγωγή που γίνεται βάσει τη ζήτηση αγοράς με συγκεκριμένα μέσα διαχείρισης. Τέλο επαναλαμβάνω και αυτό που έχω ξαναπεί και που έχουμε γκρίνει με άλλες εκθέσεις εδώ στην Επιτροπή μας. Εκθεσιντές, για παράδειγμα, για τις ποσοστώσει ζάχαρη. Νομίζω ότι πρέπει να παραταθούν τα μέτρα μέχρι το 2020 και τα δικαιώματα ε, φύτευσης αμπελιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να απαντήσει και σε κάτι άλλο. Είπατε ότι σαν μοντέλο έχετε πάρει τις οργανώσεις παραγωγών οποροκυπευτικών και αυτό το μοντέλο θέλετε να χρησιμοποιήσετε και σε άλλα προϊόντα. Όμως αν γενικευθεί έτσι το θέμα τότε υπάρχουν άρθρα το 122, 125 β και 125 τρίτο που λέει ότι το καταστατικό πρέπει να ανταποκρίνεται στις ειδικέ ε, περιπτώσεις, στις ιδιαιτερότητες. Αυτό τι σημαίνει, ότι αυτό το ειδικό τι γίνεται, γίνεται κατά εξουσιοδότηση πράξη και οι εξαιρέσεις για άλλους τομείς τι θα γίνει με αυτό. Οι, τα παροκυπευτικά πρέπει να έχουν τις εξαιρέσεις που τους πρέπουν, ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες. Σίγουρα θα συνεχίσουμε να συζητάμε αυτό το θέμα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ να απαντήσει σε ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Σα θυμίζω ότι έχουμε εκπρόσωπο τη Κομισιόν εδώ που θα μπορέσει να παρέμβει και εκείνος. Ρέιμερ τώρα. Κυρία Γαρσία πρώτα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Ταντάν για τα όσα μα είπε. Όντω είναι πολύ σημαντικό το θέμα του. Η αλήθεια είναι ότι οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φτωχέ στο θέμα τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική και τον κανονισμό ενιαία ΚΟΑ. Δεν αντιμετωπίζονται τα πιο σημαντικά προβλήματα που είναι οι αλλαγές στις τιμές και το ευάλωτο των αγορών. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα λοιπόν το οποίο να είναι πιο πρωτότυπο από αυτό που προτείνει η Επιτροπή. Δεν έχω ακούσει πάντως κάποια πράγματα σήμερα το απόγευμα, όπως είναι η νομική ασφάλεια για τους κανόνες ανταγωνιστικότητας. Είναι κάτι το οποίο λείπει από τον γεωργικό τομέα. Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές πρέπει να επιτρέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ώστε οι οργανώσεις να μπορούν να ελέγχουν την ε, εμπορία η παράληψη αυτή νομική έχει οδηγήσει σε περιπτώσεις όπως είχαμε στην Ισπανία όπου οι αρχές πήραν ε, πρωτοβουλία, στο ελαιόλαδο για παράδειγμα, να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά. Είναι μια ευκαιρία πάντως για να το λύσουμε αυτό το ζήτημα. Έπειτα, οι μηχανισμοί παρέμβασης δεν ε, πάνε γρήγορα, δεν είναι καλοί. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να το ξαναδούμε. Υπάρχουν και προβλήματα στην παραγωγή οπωροκυπευτικών, όπου όταν υπάρχει κρίση που την διαχειρίζονται οι οργανώσεις των παραγωγών, η αντιμετώπιση δεν είναι αποτελεσματική μέχρι τώρα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ταμείο, πέρα από τα λειτουργικά ταμεία, των ε, παραγωγών των κλάδων με αυτό το σκοπό. Καταστάσεις όπως είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι, με το η κόλλη είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα, τι ταμείο πρέπει να προβλέψουμε γι' αυτό. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν είναι ικανοποιητικά. Δεν μπορούν να πάρουν ε, χρήματα κάποιοι κλάδοι που θα έπρεπε και στην περίπτωση του e είδαμε ότι η διαχείριση δεν ήταν καλή. Ένα άλλο σημείο που πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον και θα έπρεπε να δούμε είναι μία λύση στις κρίσεις όπως εκείνη του ελαιόλαδου. Πρέπει τις τιμές αναφοράς να τις ξαναδούμε για την ε, ιδιωτική αποθήκευση και διαχείριση. Κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε είναι να καλύψουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν στον μηχανισμό ετοιμών εισαγωγής πριν από λίγο καιρό, εδώ στο Κοινοβούλιο, συζητήσαμε τη Συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μαρόκο και εκεί συζητήσαμε το θέμα τη τιμή τη ντομάτα. Είναι σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να ε, αποκτήσουμε ένα σύστημα που θα μας επιτρέψει, που θα επιτρέπει μάλλον στις εθνικές τελωνιακές αρχές να λάβουν υπόψη τους το θέμα αυτό των τιμών εισόδου, έτσι όπως δηλώνονται είναι κάτι που πρέπει να συμπεριλάβουμε τώρα που συζητάμε τις ενιαίες ΚΟΑ, να μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να μας ξεφύγει. Υπάρχουν και θέματα όπως είναι οι σχέσεις των βιομηχανικών ε, παραγόντων. Είναι κάτι που συζητήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών, αν δεν απατάμε. Ο κλάδος ζητάει συμβάσεις όπως το ζητά και ο γαλακτοκομικό τομέας. Το ζητάνε λοιπόν και αυτοί να υπάρχουν ε, συμβάσει λοιπόν, κάτι το οποίο θα βοηθούσε και τους παραγωγούς οποροκυπευτικών, που είναι ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι πρέπει η... βοήθεια που, οι βοήθειες που δίνονται στον γεωργικό τομέα είναι πολύ βασικές και η κυρία Λούλινγκ το έχει πει πολλές φορές μέχρι τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη γεωργία μας και πρέπει να συνεχίσουν οι ενισχύσεις αυτές να υπάρχουν. Έπειτα η δημοσιοπαρέμβαση παρέμβαση στο κρέας, χείριο, αίγιο κλπ. είναι επίσης πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αφήσουμε απ' έξω. Νομίζω ότι έχουμε πολλούς στόχους για αυτήν την ενία ΚΟΑ και καλά θα κάνουμε να τους πετύχουμε. Ευχαριστώ. Μπρίτα. Ε, Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι φαίνεται, προσπαθεί να ενσωματώσει όλη τη γεωργική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε μια μεγάλη οργάνωση αγοράς, τεράστιο έργο. Όταν μιλούμε δε για μέσα κρίση, για όργανα για την εντόση τη κρίση. Καλό θα είναι να συμφωνήσουμε τι σημαίνει κρίση. Πώ την ορίζουμε, από ποιο σημείο θεωρείτε ότι έχει εμφανιστεί μια κρίση, και πώς ε, την ε, αντιμετωπίζουμε. Ε, επί παραδείγματι έχουμε μόνο κλιματικής προελεύσεως φυσικές καταστροφές, έχουμε να κάνουμε με ιούς, όπως με τον ιό της πνευμονίας και άλλους. Δίκτυα ασφαλείας, πώς το προσδιορίζουμε και πώς το διαμορφώνουμε οι επιστροφές στις εξαγωγές σε παραδείγματι δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο περιπτώσεις κρίσεως αλλά και δυνατότητα ε, διατήρησης ενός προϊόντος ε, σε περίπτωση μεγάλης πτυτικότητας αγοράς όπως είχαμε δει με το γάλα. Ταμείο Αντιμετώπισης των Επιπτώσεων της Παγκοσμιοποίησης και επέκτασή του κατά τη γεωργία. Ε, είναι το κατάλληλο όργανο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χειρουργίας. Η δυνατότητα λογιστικά για έναν ε, γεωργό να καταθέσει μια αίτηση, να συμπεριληφθεί δηλαδή στην, ε, να υπαχθεί δηλαδή στο μέτρο του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με τι μεγάλε επιχειρήσει, τι βιομηχανικέ επιχειρήσει, είναι πάρα πολύ περιορισμένη και δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο αυτό το μέσον για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Επίσης, ίσως θα ήταν καλό για λόγους και αμοιβαιότητας να στηρίξουμε ορισμένα μέτρα ε, και να στήσουμε τη στήριξη και από τον Γεωργό. Φερρυπίν στη Γερμανία ήδη για τις επιζωτίες έχουμε προβλέψει στο σχετικό ταμείο να συμμετέχουν οι Γεωργοί οικονομικά. Αυτό είναι ένας τρόπος πιστεύω και είναι ένας τρόπος επίσης να αντιμετωπιστούν κάποιες πρώτες ζημίες, να καλυφθούν κάποιες πρώτες ζημίες, όχι βέβαια μια μεγάλη ευρεία έκτασης καταστροφή που θα μπορούσε να επιφέρει μια ε, διαδεδομένη επιζώτια στην Ευρώπη, Φέρει, Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το καλύψει μέσα από μια ασφάλιση τέτοιου τύπου. Και όταν μιλούμε για διαχείριση κρίσεων, εννοούμε ότι η Επιτροπή αλαμβάνει μόνη στην απόφαση. Συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Μπορεί με ταχεία αντίδραση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις ή χρειάζεται και το Κοινοβούλιο να την οθήσει. Και βέβαια σε αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία τι είδους συμμετοχή θα προβλεφθεί για το Κοινοβούλιο. Όταν μιλούμε δε για ενός παραγωγών, Βεβαίω θέλουμε να τι ενισχύσουμε, βεβαίω θέλουμε να έχει πιο ισχυρή διαπραγματευτική θέση ως ο Γεωργός κατά τη διαπραγματεύση του προϊόντου του, αλλά δεν πρέπει και να λησμονούμε ότι πρέπει στην περίπτωση και αυτών να ισχύει το δίκαιο το σχετικό με τον ανταγωνισμό, δηλαδή η απαγόρευση των καρτέλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Μπρίτα. Ακριβώς γι' αυτό αύριο στην συνεδρία στο συντονιστών θα μιλήσουμε για την πρόταση αυτή για να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό δρόμο. Η Ελίζαμπεθ Κόστιντζερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τον Μισελ Ντοντά για την έκθεσή του, την παρουσία της έκθεσής του. Είμαι πεπισμένη ότι τα μέσα που έχουμε τώρα στις αγορές είναι πάρα πολύ σημαντικά και αποτελούν κομμάτι και του δικτύου ασφαλείας καλό θα είναι να έχουμε επαρκή προστασία για τους γεωργούς οι οποίοι για διάφορους λόγους ε, κινδυνεύουν από εξωτερικούς παράγοντες και ιδιαίτερα στους τομείς που παρουσιάζουν θετικότητα τιμών. Υπάρχουν αρκετοί τομεί που παρουσιάζουν τεράστιε διακυμάνσει και άρα χρειάζεται και περισσότερη διαφάνεια και περισσότερο ειδικό βάρο των γεωργών στην αγορά. Αυτό είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει και με μεγαλύτερη προσοχή να παρατηρούμε, να επιοπτεύουμε την διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων. Αντίστοιχα θα πρέπει να προσαρμοστεί το δίκαιο περί ανταγωνισμού στην ε, παρουσία σε μια αγορά συγκεκριμένα ε, σε έναν τομέα και σε μια περιοχή ενός οδηγού ενδεχομένως σε κυριαρχή θέση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν χρειάζονται ειδικέ δομές. Πρέπει απλώς να βελτιώσουμε ή να προσαρμόσουμε ή να επεκτείνουμε δομές εφιστάμενες. Και αυτό με μια καλή προστασία. Ελάχιστες προδιαγραφές, μέτρα προστασίας που θα προστατεύουν και ε, τον παραγωγό από μεγάλες διακυμάνσεις τιμών. Για δε την αγορά γάλακτος πολύ σύντομα, μια και πρόσφατα εγκρίναμε τη σχετική έκθεση στην αγορά, στην Ολομέλεια θα ήθελα να επισημάνω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο, για ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα που θα χρειαζόταν οπωσδήποτε να έχουμε από το 2015 και μετά χρειάζεται να τεθεί σε εφαρμογή και νομίζω ότι με την έκθεση αυτή το Κοινοβούλιο αποστέλει και γι' αυτό ευχαριστώ και τους συντάκτες εκθέσεως σαφές μήνυμα για την αδύναμη σχέση στην οποία βρίσκονται οι παραγωγοί γάλακτος στην αλυσίδα του προϊόντος. Και ίσως θα πρέπει να διαρωτηθούμε κατά πόσον ε, ορισμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να καταβάλουν σημαντικές κυρώσεις ή ποινικέ ρήτρες για τον τομέα του γάλακτος, ενώ κάποια, άλλη δεν, κάποια άλλα δεν χρειάζονται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει εμείς να δώσουμε τον τόνο και να αναλάβουμε τις σχετικές πρωτοβουλίες. Ε, Επίση, περιοχές με μειονεκτήματα λόγω γεωγραφικής ε, θέσης ε, ή διαμόρφωσης ε, θα πρέπει βεβαίως να τα αντιμετωπίσουμε μια ιδιαίτερη φροντίδα και μέρημνα. Για την αγορά σακχάρεως και την ποσόστοση που εκπνέει το 2020, θα ήθελα να παραδέψω στην έκθεση που έρχεται μόλις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πω ότι έχουμε πει ρητά πως θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η ποσόστοση μετά το 2020. στην ε, μελέτη επιπτώσεων, στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουμε ότι δεν ε, μπορεί κανείς να προβλέψει ε, τα στοιχεία και τα ποσοστά τα οποία θα ισχύουν μετά το 2020, παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει συμπεριλάβει στο κείμενό της και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ε, προβλέψουμε ενδεχομένως διαφορετικές συνθήκες για τον τομέα της ζάχαρης μετά το 2020. Και ανάλογα θα πρέπει να ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις με κύριο στόχο, με πρωταρχικό στόχο στην Ευρώπη εν γέννη να εξασφαλίσουμε την αυτονομία σε τρόφιμα, ώστε να μην χρειάζεται να εξαρτώμεθα από εισαγωγές. Άρα το ζήτημα της ποσότητας της σάχαρης και του τρόπου με τον οποίο θα χειριστούμε το θέμα αυτό έχει τεράστια σημασία. Ο κύριος Μποβέ και μετά Μακίνες. Euh, Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Μισελ Νταντά για τη δουλειά του. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του, λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση στην οποία θα βρισκόμαστε σε λίγο καιρό, τότε που θα λέμε τι έκανε η Ευρώπη και τελικά βρίσκεται συνέχεια σε κρίση. Αυτό που προσπαθεί να οργανώσει η Επιτροπή, η Επιτροπή και όχι το Κοινοβούλιο, πρέπει να έχει υπόψη το εξή. Όταν διαλύουμε ε, τις δομές, θα υπάρξει ανισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά. Αν όλοι οι αγρότες σκέφτονται το ίδιο πράγμα συγχρόνως, έχουμε υπερπαραγωγή και άρα καταστροφή. Ναι, είμαστε σε κρίση. Άρα το πραγματικό ερώτημα τώρα είναι, με αυτή την ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει όλα, όλους τους μηχανισμούς ε, ισορροπίας ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά, αυτό το θέμα της αποθήκευσης θα βοηθήσει. Εδώ είναι το πρόβλημα ουσίας και γι' αυτό εύχομαι καλό κουράγιο στον Μισελ το θέμα και δεν θα μπούμε τώρα στο θέμα κρασί ή ζάχαρη, αν και είναι ενδιαφέρον να μιλάμε για το κρασί. Υπάρχει μια συνάντηση του αμπελονικού τομέα σήμερα το βράδυ. Αν λοιπόν κάνουμε όπως θέλει η Επιτροπή, δηλαδή εγκαταλείψουμε τα δικαιώματα στη φύτευση, τότε μπαίνουμε σε μια πλήρη αναρχία και θα είναι η έκρηξη και του όγκου κάπου και αλλού δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να προχωρήσουν και θα έχουμε κρίση. Ε, τι θα κάνουμε λοιπόν με αυτό. Εντάξει, εδώ θα σταματήσω, δεν θέλω να πω πολλά επί της ουσίας. Πιστεύω όμως ότι πραγματικά το πρόβλημα έχει να κάνει με τον όγκο ζήτησης και προσφοράς Ξανασκεφτείτε το σας παρακαλώ, γιατί αυτό που κάναμε για το γάλα δεν άλλαξε σε τίποτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ονομασίες προέλευσης. Με το ζόρι δέχτηκαν κάποια εξαίρεση. Είναι απαράδεκτο. Δεύτερον, τι κάνουμε με το κόστος παραγωγής ε, των γεωργών στον ορισμό των τιμών. Σήμερα οι αγρότες έχουν ε, τεράστιο, τεράστιες διαπάνες, τεράστιο κόστος. Έκανα πριν από μερικούς μήνες μια έκθεση που ψηφίστηκε σήμερα. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αγρότες καθόλου οι δικές τους οι δαπάνες. Πώς θα το συμπεριλάβουμε όμως για να μπορούν να τίθενται σε εφαρμογή οι κατάλληλοι μηχανισμοί. Τέλος, πολύ σωστά θα γίνει η συζήτηση και ελπίζω αύριο το πρωί οι συντονιστές να δουλέψουν ε, καλά πάνω σε αυτό το ταμείο για τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Αυτή είναι μια μεγάλη παγίδα που έχει μπει στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να δεχτούν το ταμείο αυτό ε, προσαρμογής. Είναι σήμερα σαν να μας ε, ζητούν να ετοιμάσουμε τη θηλιά για να κραμαστούμε οι ίδιοι. Μα είναι μαζοχισμός. Πάνω σε αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όπως και στην πρώτη συζήτηση, η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να απορρίψει και πάλι απόλυτα το Ταμείο αυτό προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση για τον γεωργικό τομέα. Είναι κάτι που στρίβει την πλάτη σε κάθε γεωργική πολιτική. Μια για πάντα. Είναι σαν να λέμε ότι τελικά δεν αποφασίζεται εδώ στις Βρυξέλλες η γεωργική πολιτική, αλλά στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη Γενέβη. Μάλιστα, αυτό το θέμα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης μας ε, ανησυχεί όλους και μας ενδιαφέρει όλους. Θα πρέπει να αποφασίσουμε και αύριο θα γίνει ad hoc συνεδρίαση των συντονιστών για αυτό το θέμα. Μαγκίνες και μετά Πατράων σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί οι συνάδελφοι κάλυψαν διάφορα θέματα. Ευχαριστώ καταρχήν τον Μισελ ε, Νταντά για την παρουσίασή του και θα ήθελα να σας ζητήσω να ασχοληθείτε πιο άμεσα γιατί καταλαβαίνω πως σωστά εστιάζουμε στις άμεσες πληρωμές αλλά ίσως οι ομάδες πίεσης να μην προσέχουν αρκετά τα μέτρα για την αγορά και όταν έχουμε μια κρίση μετά θα αναρωτιόμαστε γιατί συνέβη αυτό. Γι' αυτό και συμφωνώ με τη γενική συζήτηση για την ε, μεταρρύθμιση της κοινή γενική πολιτικής. Ε, ε, το θέμα είναι... Μισελ, αν μπορείς κάπως να μας εξηγήσεις κάπως περισσότερο το πώς θα μπορεί να ενεργήσει γρήγορα η Επιτροπή ε, με βάση ένα κατώτατο όριο. Το θέμα των ε, ενώσεων παραγωγών ανατομέα, νομίζω πως ε, η Κομισιόν βασίζεται σε αυτό για την αύξηση της ε, δύναμης των παραγωγών και το στηρίζω. Νομίζω υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή με την ε, λειτουργία κάποιων οργανώσεων ε, παραγωγών. Πρέπει να εξετάσουμε πώς λειτουργούν και πώς θα μπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Επίσης θα ήθελα το Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη το τι γίνεται παράλληλα στην Κομισιόν με την ομάδα υψηλού επίπεδου για την λειτουργία της αλυσίδα παροχής τροφίμων Πράγμα από το οποίο θα πρέπει νομίζω να, να αντικατοπτρίζεται και στις συζητήσεις μας εδώ, γιατί μιλάμε για το ίδιο θέμα. Αλλά το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στη συζήτηση που γίνεται στην Κομισιόν στην ομάδα επιπέδου. Το θέμα είναι πως όταν κάτι πάει στραβά θα πρέπει να έχουμε αρκετά μέτρα τα οποία να χρησιμοποιήσουμε γρήγορα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κρίση. Στον τομέα του γάλακτος ήμασταν αργοί, μη αποτελεσματικοί και οι κτηνοτρόφοι πέφεραν. Με αυτή την ΚΟΑ πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιου είδου προβλήματα. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σου, Μισελ. Σα ευχαριστώ. Α, ναι, και να μην χάσω, ξεχάσω και να υποστηρίξω, Πρόεδρε, τα σχόλια της κυρίας Κόστιγκερ σε σχέση με την κατάσταση των ποσοτώσεων του γάλακτος. Για κάποια κράτη μέλη δεν υπάρχει ομαλή προσγείωση και χρειάζεται η Κομισιόν τουλάχιστον να αρχίσει να εξετάζει την κατάσταση και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα για τα κράτη μέλη όπου υπάρχει ζήτημα τέτοιο. Και σίγουρα εγώ τον υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μαρία. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης της κρίσης της αγοράς ε, που το έχουμε συζητήσει επανειλημμένω και είναι ευθύνη ολόκληρη τη Επιτροπή. Πρέπει να δουλέψουμε και να στηρίξουμε τη δουλειά του Νταν Τεν και όλων των σκιωδών εισηγητών, ώστε να φτάσουμε σε μια πρόταση που να δώσει τι απαντήσει που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Η πατράου Νέβες και μετά κλείνει ο Τζιμ Νίκολσον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί ήθελα απλά να τονίσω δύο πτυχές. Η μία σχετίζεται με την οργάνωση μέτρων επίγουσας ανάγκης που πάντα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ισότητας. Εάν δεν είναι δυνατόν να θεσπιστούν κάποια ε, υποχρεωτικά ελάχιστα όρια για όλα τα κρατη θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πολύ διαφορετικές καταστάσεις σε όλα τα κρατημέλη και ανάμεσα στους Ευρωπαίους Γεωργούς. Αυτή τη στιγμή που θέλουμε να, να οργανώσουμε μια κοινή γεωργική πολιτική και βλέπουμε ότι θέλουμε να είμαστε πιο, πιο μεγάλες είναι οι αγορές και η ανταγωνιστικότητα είναι το μεγάλος αγώνας. Πώς θα κερδίσουμε σε αυτό το επίπεδο και πώς θα είναι δίκαιος αυτός ο αγώνας εάν δεν υπάρχει μια ελάχιστη κοινή πλατφόρμα Πριν από λίγο είπα ότι η Πορτογαλία και η Ισπανία περνούν μια κατάσταση δραματική, επικρατεί τρομερή ξηρασία και είναι αλήθεια ότι οι Πορτογάλοι γεωργοί δεν έχουν δυνατότητα να ασφαλιστούν κατά της ξηρασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν υπάρχει δυνατότητα ε, και ο καθένας ε, πρέπει να δεχτεί τις ε, συνέπειες. Ενώ οι γείτονες, οι Ισπανοί, μπορούν να ασφαλιστούν κατά της εξηρασίας. Βλέπετε ότι το σύνορο υπάρχει λοιπόν και η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από τη μια χώρα στην άλλη. Χρειάζεται λοιπόν σε τέτοια μέτρα επίγουσες ανάγκες να υπάρχουν κάποια ελάχιστα υποχρεωτικά μέτρα, όρια, γιατί διαφορετικά δεν θα είναι δυνατόν να έχουμε μια γεωργική πολιτική τέτοια όπου η ανταγωνιστικότητα να είναι ο γνώμονας για τους γεωργούς. Δεύτερη πτυχή είναι ο τομέας του γάλακτος, όπως ε, θα φανταζόσασταν. Να σας θυμίσω, ως όλους τους αγαπητούς συναδέλφους, ότι η έκθεση που εγκρίναμε για τις συμβατικές σχέσεις δεν αντικαθιστά τις ε, γαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Είναι ένας μηχανισμός ρύθμισης και ενημέρωσης για την αγορά αυτές οι ποσοστώσεις και που δεν επιτρέπεται πια. Και βλέπουμε ότι αυτό το έγγραφο για το πακέτο για το γάλα δεν λαμβάνει υπόψη τους συνεταιρισμούς. Ξέρουμε πως υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί. Βλέπουμε επίσης πως η έννοια του συνεταιρισμού διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και εκτός από όλα αυτά έχουμε και περιοχές μειονεκτούσες που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από την γαλακτοκομική παραγωγή και με μια τελείως απελευθερωμένη αγορά δεν υπάρχει καμιά εγγύηση πως αυτές οι περιοχές θα συνεχίσουν να παράγουν ε, γάλα και τα, οι επιπτώσεις της έλλειψης παραγωγής γάλακτος σε αυτές τις περιοχές θα είναι καταστροφικές όσον αφορά τον πληθυσμό, τη χωροταξία και την φροντίδα και τη συντήρηση της ίδιας της περιοχής κάθε φορά. Ακόμα μια πτυχή όσον αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τα γεωργικά θέματα, όπως αναφέρθηκε ήδη. Ήρθε αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας και εγώ είπα ότι πρόκειται για ένα δηλητηριασμένο δώρο Θα πρέπει ωστόσο να το συζητήσουμε για να δούμε ποια θα είναι η κοινή θέση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η Κομισιόν να απεκτηθεί των ευθυνών της σε σχέση με τα όσα θα έπρεπε να κάνει για την προστασία της γεωργίας και όχι για τη χρήση της γεωργίας ως αντάλλαγμα. Σας ευχαριστούμε. Ο Τζιμ Νίκολσον. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα υποστηρίξω τον κύριο Ντόντα και την προσέγγιση στο θέμα. Αν και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Ένα πράγμα που μας έμαθε η κρίση είναι ότι υπάρχει ανάγκη για παρέμβαση υπάρχει ανάγκη για δίκτυα ασφαλείας. Σε ποιο επίπεδο, με ποια ταχύτητα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αυτό το δίκτυο ασφαλείας, στον ένα τομέα ή στον άλλον, αν εμφανιστεί η κρίση. Όλα αυτά είναι απαντήσεις που καλούμε να δώσουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ε, λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά πάντως, εάν αποφασίσουν οι γεωργοί να παράγουν περισσότερες, μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι μπορεί να απορροφήσει η αγορά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί δεν νομίζω ότι ο φορολογούμενος της Ευρώπης είναι διτηθειμένος να επανέλθει στο φαινόμενο των ε, όρεων βουτύρου και λιμνών ε, γάλακτος που είχαμε στο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν περάσει πια. Και έτσι πρέπει να βρούμε έναν ρόλο και ένα μηχανισμό ε, λειτουργίας αυτού του δικτύου ασφαλείας ε, ικανοποιητικό και πολύ καλά σταθμισμένο. Αυτές οι ε, ενός παραγωγών και διατομιακές μάλιστα πρέπει να τις κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί ένα απολύτως ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς περιθώριο κάποιο κράτος μέλος να ε, προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα ή επιδότηση. Δηλαδή το common κοινό από την κοινή γεωργική πολιτική να μείνει, να μην χαθεί η λέξη κοινό, κοινή γεωργική πολιτική. Και πρέπει βεβαίως να πείσουμε και τους γεωργούς μας ότι ναι, μπορεί να υπάρχει κάπου κάποιο μικρό πλεονέκτημα για κάποιον υπό ορισμένε συνθήκες, αλλά αυτό είναι πάντοτε ε, περιορισμένο στο χρόνο, βραχυπρόθεσμο δηλαδή, και περιορισμένο και σε έκταση. Και ότι εν γέννη η γεωργική πολιτική είναι αυτή που προσφέρει τα μέγιστα πλεονεκτήματα για τους πάντε. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Ντοντά ότι θα πρέπει να μην χαθεί ο, ο ρόλος του ε, γεωργού, και χωρίς να γνωρίζω θέματα δημοσιονομικά, θέματα του προϋπολογισμού, ε, εάν δεν έχει αρκετή χρηματοδότηση το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, νομίζω ότι έχει κανένα ρόλο να διαδραματίζει. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να επαναλάβω στον αδέλφο να πω και νωρίτερα ότι εάν κανείς πάει να παραγάγει κάτι, ε, ένα προϊόν για το οποίο δεν υπάρχει αγορά, πολύ προσοχή χρειάζεται, διότι κάποια στιγμή θα πει ο, ο καταναλωτής, θα πει ο πολίτης, φτάνει πια, δεν θέλουμε άλλο. Ευχαριστώ κύριο Σικέρσκι. Πρόεδρε, πολύ συχνά μιλώ για τις γεωργικές αγορές που δεν είναι σε θέση να, να ε, επιλύσουν τα προβλήματα της αγοράς της προσφοράς καλύτερα που προξενούν Γιατί υπάρχει πάντα μια κάποια ε, πτυτικότητα των αγορών στον το γεωργικό τομέα. Πτυτικότητα που εξαρτάται από τις κλιματικές ε, εξελίξεις, Φερρυπίν, από τις κλιματικές συνθήκες δηλαδή. Επίσης ε, από τις μεγάλες διαφορές μεταξύ μεγάλου και μικρότερου παραγωγού. Και άρα δεν μπορούμε να έχουμε μία ενιαία και συνεπή προσέγγιση στην αλυσίδα της παραγωγής. Όλες αυτές λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται Και νομίζω ότι οι προτάσεις για τις ευρωπαϊκές αγορές που εξετάζουμε δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματά μας. Και έτσι οι γεωργικές αγορές κινδυνεύουν να επαφεθούν τελείως στην δύναμη, στις δυνάμεις της αγοράς. Να μην υπάρχει κανένας έλεγχος δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλα αυτά που έφτασαν με καθυστέρηση, όλα αυτά μέτρα που δεν ε, ε, λήφθησαν εγκαίρως, οδήγησαν τελικά σε πολύ πιο υψηλό κόστος. Και εάν δεν μπορέσουμε να στηρίξουμε τους ε, μικτούς αυτούς ε, οργανισμούς, μικτές αυτές ενώσεις ε, των ε, παραγωγών, θα πρέπει να περιμένουμε πολύ πιο υψηλό κόστος για τα γεωργικά τρόφιμα από το χωράφι μέχρι το πιάτο μας. Όταν μιλούμε για οργάνωση, κοινή οργάνωση αγοράς, πολλά πράγματα εννοούμε και ξέρω ότι οι διαπραγματεύσεις στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου συνεπάγονται κόστος για τον Γεωργό υψηλό για το οποίο θα πρέπει να τον αποζημιώσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σιγέρσκη. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν, στον ε, Διευθυντή Φεστάιλεν και μετά στον εισηγητή για να ολοκληρώσει τη συζήτηση του θέματος. Παρακαλώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πιστεύουμε πως οι προτάσεις που έχουμε αποβάλει στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ για μετά το 2013 τοποθετούνται στη λογική των διαφόρων ε, ε, ρυθμίσεων που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, από το 1992 και ε, στη συνέχεια. Εμείς ε, στηρίζουμε το εισόδημα βασικά. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο έχουμε γίνει πολύ ανταγωνιστικοί θα έλεγα. Αν δείτε την κατάστασή μας για τα πιο σημαντικά προϊόντα όσον αφορά τις τιμές σε σύγκριση με την παγκόσμια αγορά, είμαστε ανταγωνιστικοί. Αν δούμε τα δημητριακά για το σιτάρι και το κρυθάρι, οι τιμές είναι παρόμοιες με τους κύριους ανταγωνιστές μας και αυτό σημαίνει πως είμαστε ε, καθαροί εξαγωγής χωρίς επιστροφές. Ε, και στον γάλα έχουμε το ίδιο, εξάγουμε χωρίς ε, αποζημιώσεις στις εξαγωγές και το τυρί και το βούτυρο γίνεται χωρίς επιστροφές. Αν δούμε το τομέα της ζάχαρης που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ε, πολύ χαμηλή η τιμή σε σχέση με την εσωτερική μας τιμή, είδαμε τον τελευταίο χρόνο ότι παγκοσμίως η τιμή της ζάχαρης ήταν ακόμη ψηρότερη. Υπάρχει μια μεγάλη μετατροπή από τη μια πλευρά της εσωτερικής μας τιμής, των ιστορικών μας τιμών μάλλον και των εξωτερικών τιμών. Και αυτό φυσικά οφείλεται στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγορές αλλά και στην λογική των μεταρρυθμίσεών μας. Έχουμε λοιπόν τώρα κάποια επίπεδα ασφαλείας που είναι το αποτέλεσμα αυτών των μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια των ετών, εξακολουθούν να ισχύουν και στον τομέα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, στον τομέα του γάλακτος, λειτουργήσε πολύ καλά το σύστημα. Παρενέβημεν και βάλαμε και ένα κατώτατο όριο στην αγορά. Το ίδιο λοιπόν θα να χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον, καθώς και ιδιωτική αποθήκευση και παρέμβαση. Τώρα βέβαια το θέμα είναι, θέλουμε να αυξήσουμε αυτό το δίκτυο ασφαλείας, ναι ή όχι. Και το θέμα προκύπτει ας πούμε για το, τα τρόφιμα και τα προκυπευτικά. Είναι λεπτό το ζήτημα κύριε Πρόεδρε αυτό, γιατί κάναμε τόση δουλειά για να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα πρέπει να προσέξουμε να μην χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην παγκόσμια αγορά. Ένα άλλο τομέα που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ένα παράγοντα μάλλον, είναι ότι αν τώρα δείτε τις προτάσεις μας, έχουμε βεβαίως μετατρέψει τον προϋπολογισμό από στήριξη της αγοράς 100% στο 95% άμεση στήριξη εισοδήματος. Και υπάρχουν λίγα χρήματα που έχουν μείνει για την στήριξη της αγοράς. Αν θυμάμαι καλά ήταν ε, 2,7 δις ευρώ είναι μέχρι το 2015 και ένα σημαντικό τμήμα αυτού είναι για το κρασί και για τα τρόφιμα και απορροκυπευτικά. Ε, και η πρότασή μας είναι να επεκταθούν οι άμεσες πληρωμές και στα τρόφιμα και απορροκυπευτικά που δεν χαίρουν των άμεσων πληρωμών αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν ο τομέας αυτός ε, έχει τύχει πολύ καλής μεταχείρισης κατά τη γνώμη μου. Τώρα όσον αφορά το Ταμείο Κρίσης. Θα έλεγα ότι τα τρία άρθρα που στηρίζουν αυτό το ταμείο είναι αποτέλεσμα εμπειριών ετών όπου έχουμε φτιάξει τη νομική βάση για να παρέμβουμε σε περίπτωση κρίσης για τους μεμονωμένους τομείς και έχουμε επεκτείνει αυτές τις νομικές βάσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς. Αυτούς δηλαδή που για την ώρα, αυτοί που εξαιρούνται μάλλον για την ώρα είναι η πατάτα και το κρέας ε, αλόγου. Αλλά δεν έχουμε ποτέ παρέμβει σε αυτούς τους τομείς. για το Ταμείο Κρίσης. Τι είναι η κρίση, ρώτησαν διάφοροι ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να προσέξουμε για να ορίσουμε μια τέτοια κρίση, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει μια κρίση και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω μεγάλη ευελιξία από την πλευρά της Κομισιόν για να μπορούμε να παρέμβουμε σε μια κρίση και να μην περιοριζόμεθα από έναν ορισμό που δεν καλύπτει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, και κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι ότι ως Κοινοβούλιο επίσης συμμετέχετε στην εκτέλεση του Ταμείου της Κρίσης. Αυτό εσείς πρέπει να συμφωνήσετε για την ε, απελευθέρωση των κονδυλίων και φυσικά σε μια κρίση θα πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και γι' αυτό θα σας ζητήσουμε να προχωρήσετε στο πλαίσιο μιας ε, ταχείας διαδικασίας, fast track procedure, όπως γίνεται ας πούμε και για την βοήθεια σε επίγουσα κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τη ζάχαρη και το κρασί, τον νίνο ήδη έχουμε συζητήσει νωρίτερα τη ζάχαρη και είπα ότι η εσωτερική ζάχαρη έχει γίνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και σας έδωσα και παράδειγμα. Έχουμε την εντύπωση, αν, αν δείτε καθημερινή διαχείριση της αγοράς ζάχαρης όπως αυτή γίνεται από την ε, Κομισιόν, δεν περιορίζουμε απαραίτητο στην εσωτερική μας παραγωγή στο να ε, αποφελούνται δυνατότητες σε διεθνές επίπεδο, διότι εξακολουθούμε να ακολουθούμε το πάνελ του ΠΟΕ Έχουμε ακόμη περιορισμούς για το πού μπορούμε να πουλήσουμε την ζάχαρή μας. Και αφού είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί να, χρησιμο... γιατί να εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτούς τους περιορισμούς. Και τα δικαιώματα τώρα φύτευσης. Υπήρχε μια άποψη ότι αν καταργηθούν αυτά, θα υπάρξει μια έκρηξη παραγωγής ε, ίνου. Να σας θυμίσω, αν μου επιτρέπετε, ότι τα δικαιώματα φύτευσης δεν είναι όπως οι ποσοστώσεις ε, γάλακτος ένας μηχανισμός ελέγχου όγκου. Είναι ένας μηχανισμός που αποφασίζει ποιος παράγει, αλλά μετά ο μεμονωμένος παραγωγός αποφασίζει ποιος είναι ο όγκος που θα παράγει ένα εκτάριο. Είναι κάπως διαφορετικό το σύστημα, αρκετά διαφορετικό το σύστημα κύριε Πρόεδρε. Τώρα, αν ε, δούμε τώρα τις ε, ενώσεις παραγωγών. Όπως ξέρετε έχουμε προτείνει την επέκταση των ενώσεων παραγωγών σε όλους τους τομείς και πρόκειψε το θέμα του κατά πόσο πρέπει να ακολουθήσουμε το πρότυπο του γάλακτος, το οποίο προέκυψε σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις όπου φεύγουμε από τις ποσοστώσεις και ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο συζητήθηκε μέσω διαπροπατεύσεων. Αν δεχτούμε αυτό το μοντέλο όσον αφορά το, κανόν, το δίκαιο ανταγωνισμού, χρειάζεται μια ειδική εξαίρεση. Μια ειδική εξαίρεση είχαμε για το γάλα και όπως θα θυμάστε τώρα έχουμε τη δυνατότητα οι ενώσει παραγωγών να διαπραγματεύονται το 33% του εθνική παραγωγής, αλλά δεν έχουμε τέτοιες εξαιρέσεις για τις, ενώσεις, για τις φυσιολογικές ενώσεις παραγωγών. Και όπως σας είπα το γάλα είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Τώρα, τα όσα είπε η κυρία Γκαρσία για το άρθρο 25 ABC, το οποίο έχει φύγει από την πρότασή μας και σε ποιο βαθμό έχει γίνει αυτό. Τα άρθρα αυτά αφορούν τις δραστηριότητε των ΚΟΑ και φυσικά θα τα δεχτούμε υπό ε, πράξεις κατ' εξουσιοδότηση για να είμαστε πιο ευόλεκτοι γιατί αν το τοποθετήσουμε στο βασικό κανονισμό αν θέλουμε μετά να αλλάξουμε πρέπει να περάσουμε ολόκληρη την νομοθετική διαδικασία πράγμα που μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρο. Όσον αφορά τις ε, αγορές ο κύριος Νίκολσον ζήτησε ισότιμο πεδίο για όλους τους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε τα κάτι μπελ να δώσουν τις ερμηνείες τους, πράγμα που θα οδηγήσει σε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Νομίζω πως ο τρόπος με τον οποίο διατυπώσαμε την πρότασή μας δίνει την εξασφάλιση ότι αυτές οι καταστάσεις θα αποφευχθούν. Επίσης έγινε αναφορά στην οργάνωση για τα φρούτα και απορροκυπευτικά. Δεν έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση, αλλά ο Επίτροπο Τσόλο έχει σκοπεύει να το βάλει νωρίτερα την έκθεση που, που είχαμε ε, να φτιάξουμε για το τέλος το 2013, να φτιάξει μια έκθεση λοιπόν και μελέτη αντικτύπου για τις προτάσεις αυτές. Θέλει να επιταχύνουμε δηλαδή για το προβληματισμό για τα φρούτα και οποροκυπευτικά. Επίσης έγινε λόγος για καλύτερη ανείχνευση των εισαγωγών και των τιμολογίων. Θα γίνει σχετική πρόταση στην Επιτροπή Διαχείρισης στη Διαχειριστική Επιτροπή πολύ σύντομα, ώστε να έχουμε όντως καλύτερη ανείχνευσιμότητα. Και για την ε, στήριξη, για τις μέλησες δεν αλλάζουμε κάτι. Δανεισμός για το γάλα το έχουμε συζητήσει στο πακέτο γάλακτος αυτό αν θυμάστε. Ε, δεν υπάρχει στήριξη για κάτι τέτοιο στο Συμβούλιο ώστε να ανασταλεί η συμφωνία για τις ποσοστώσεις. Είμαστε ήδη στα μέσα σχεδόν του 2012, οπότε δεν πιστεύω πως αυτή τη φάση της εφαρμογής του γάλακτος και την ομαλή προσγείωση θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως κάλυψα πάνω κάτω όλα τα θέματα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον ε, Διευθυντή Βερσλάινεν. Αφού ακούσαμε την Κομισιόν, συγχαίρω ακόμη περισσότερο τον Μισελ Νταντέν και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους και όλες που πήραν το λόγο. Όσα ακούσαμε επιβεβαιώνουν την εντύπωση που είχα σχηματίσει από τις επαφές που είχα ατομικά με τον καθένα από εσά. Ότι δηλαδή υπάρχει κάποια συνένεση. Τι βγαίνει. Βγαίνει ότι όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια κατεύθυνση συγκεκριμένη, αλλά να βρούμε τα μέσα. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό, πρώτα απ' όλα με τη γνώση, γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει στις αγορές. Και αυτό είναι που πρέπει να προσθεθεί στην πρόταση. Πολλές φορές αναφερθήκαμε στο θέμα των βαρών που επομίζονται οι αγρότες. Υπάρχει το άρθρο 17 που μιλάει για την ιδιωτική αποθήκευση και που για πρώτη φορά λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση του τομέα και όχι μόνο για τα φρούτα. Πρέπει βέβαια να αποφασίσουμε η διάταξη αυτή πρέπει να διευρυνθεί και στην ε, δημόσια παρέμβαση. Μπορεί να υπάρξει δημόσια παρέμβαση όταν οι δαπάνες αυξάνονται ακόμα και αν οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές. Έπειτα, πολλοί άλλοι αναφέρθηκαν στα οικονομικά μέσα. Πού θα βρούμε τα χρήματα αυτά, λένε. Θα τα βρούμε στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, θα τα βρούμε στο Ταμείο Κρίσης, πού. Έχουμε όμως ήδη κάποια νομικά μέσα στη διάθεσή μας και που θα έπρεπε να διευκρινιστούν παρετέρω στο κείμενο. Τέτοια μέσα παρέμβασης επιτρέπουν να μεταφέρουμε ε, χρήματα μέσα σε τρεις δομάδες κατά τη διάρκεια των οποίων το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λένε τη γνώμη τους. Όμως είμαστε ορισμένοι εδώ μέσα που συμμετέχουμε στην ομάδα εργασίας που θα δουλέψει πάνω στις δημοσιονομικές προοπτικές και το νέο τεχνικό πλαίσιο χρηματοδότησης. Ο συνάδελφος δηλαδή δεν είναι πια στην αίθουσα, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε. Μπορούμε να βγούμε από την αρχή ε, της ετήσιας διάστασης των πιστώσεων. Πρέπει δηλαδή να βρούμε έναν τύπο με την Επιτροπή Προπολογισμών που θα μας επέτρεπε σε τρία χρόνια να διατηρούμε τις πιστώσεις και να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Δεν λέω επάπειρο, λέω να τις διατηρήσουμε για παράδειγμα τρία χρόνια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα μαξιλάρι ασφάλειας. Οπότε στα πλαίσια του συνολικού ποσού να έχουμε ένα ποσό στη διάθεσή μας, αντί να προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε κάποιο άλλο με έναν άλλο τρόπο που να μην είναι τόσο καλός ε, όπως αυτά που έχουμε τώρα. Τώρα, όσον αφορά τον ορισμό της κρίσης, άκουσα διάφορες απόψεις. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει το Κοινοβούλιο να προσπαθήσει να ορίσει το ότι είναι κρίση, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε όλες τις περιπτώσεις, συνάδελφοι. Και όταν θα έχουμε καταλήξει σε έναν ε, ορισμό, να ξέρετε ότι οι νομικοί με τους οικονομολόγους θα διαφωνήσουν μεταξύ τους και ο καθένας θα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει σαν άλλο αυτή τον ορισμό του άλλου. Μην ορίσουμε λοιπόν το ότι είναι κρίση. Αντίθετα, να βρούμε τον μηχανισμό εκείνων που θα μας βοηθήσει να έχουμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή την απόφαση για το κατά πόσο πρόκειται ή δεν πρόκειται για κρίση κάθε στιγμή που θα τους ζητήσουμε να το κάνουν δηλαδή, αντί να έχουμε έναν οικουμενικό ορισμό της κρίσης που δεν θα μας πάει μακριά. Ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε πολύ. Νταντέν. Σας ευχαριστώ όλους. Και έτσι πάμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχουμε για σήμερα, που είναι το σημείο 5 και είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων. Η συγγήτρια είναι η Μαρίτ Πάλσεν, αντιπρόεδρος Πόλσεν. Σας υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή στις 19 Ιανουαρίου ενέκρινε μια δεύτερη στρατηγική για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων που προτείνει ένα σχέδιο της Επιτροπής για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Προβλέπεται ένα απλοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για την καλή μεταχείριση των ζών που πρέπει να στηρίξουν τα κράτη-μέλη για να βελτιωθούν ευρωπαϊκές προδιαγραφές και στηρίζει την διεθνή συνεργασία και θέλει οι καταναλωτές να έχουν όλες τις πληροφορίες ε, που υπάρχουν ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή ε, γραμμή. Έχουμε εδώ και εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε μπορούν και να παρέμουν. Αλλά προς το παρόν η συγγήτρια. Μάριτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώντας, ήθελα να πω ότι συνομίλησα με οποιονδήποτε είχε εκδηλώσει οδήποτε ενδιαφέρον για την προστασία των ζώων. Η βασική αρχή πάνω στην οποία επεξεργάστηκα το κείμενό μου είναι ότι το 95% των ζώων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκουν σε γεωργούς και άρα η μεταχείριση τους ξέρετε από αυτούς. Δηλαδή μιλούμε ε, για την καθημερινή εμπειρία των γεωργών. Αυτή έχει σημασία όταν συζητούμε την ευημερία των ζώων. Και Βασικά δεν προσπαθώ να προχωρήσω, να προωθήσω νέα νομοθεσία η οποία θα γεννούσε περισσότερα ακόμα επίπεδα γραφειοκρατίας και θα περίπλακε, θα περίπλακε ακόμα περισσότερο τη ζωή για τον Γιώργο. Διότι Επιβάλλονται τόσε πολλέ δεσμεύσει, υποχρεώσει για τη βιοπικιλότητα, το περιβάλλον, την ευημερία των ζώων στον γεργό, που θα πρέπει ίσως να βρούμε μια ολιστική προσέγγιση. Και να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία, οι διατάξεις, οτιδήποτε ισχύει, εν γέννη είναι σαφές και ξεκάθαρο και ε, ευχερός εφαρμόσιμο. σε αυτή τη στιγμή ε, επικρατεί το απόλυτο χάος στον χώρο της νομοθεσίας για τα ε, γεωργίες και ιδιαίτερα στον τομέα αυτών, μιλούμε για τελείως διαφορετικά σημεία, 23 διαφορετικά νομοθετήματα που μπορείτε απλούστατα να πολλαπλασιάσετε επί 27 κράτη-μέλη, διότι το κάθε κράτος μέλος ερμηνεύει το κάθε νομοθέτημα με το δικό του τρόπο για να βγάλετε το γινόμενο. Και βέβαια ο τελευταίος τροχός της αμάξης είναι μόνο ο Γεωργός, γιατί εκείνος πάλι βρίσκεται ε, καλούμενος να υλοποιήσει την ομοθεσία. είτε πρόκειται για κάποια μεγάλη γεωργική εκμετάλλευση, δεν πρόκειται για τον ε, γιδοβοσκό στο τελευταίο χωριό που έχει μόνο δεκαγίδια. Αυτό λοιπόν ε, μας υποχρεώνει να αναλογιστούμε ένα νέο τρόπο, ένα νέο σχεδιασμό, και έτσι υιοθετήσαμε το Μάιο του 2010 μια έκθεση πρωτοβουλίας που σημαίνει ότι οτιδήποτε συζητούμε τώρα θα πρέπει να ε, στηρίζεται σε απλά επαληθεύσιμα επιστημονικά δεδομένα και την ε, επαλήθευση αυτών. Και γιατί επιμένω τόσο πολύ σε μια τόσο σε μια προσέγγιση στηριζόμενη στην πρακτική και την απόδειξη των, της θεωρίας. Γιατί ακούσατε η ευημερία των ζώων είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε από τη μια όλους αυτούς που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ζώων, που ε, βροντοφωνάζουν και ζητούν περισσότερη φροντίδα και προστασία για τα ζώα, ενώ από την άλλη, στο άλλο άκρο μάλλον του φάσματος, υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι τα ζώα δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια μηχανία, από ένα μηχάνημα. Και ως εκ τούτου πρέπει να συγκεράσουμε τις δύο, τα δύο αυτά άκρα και να βρούμε μια χρυσή τομή, μια μέση οδό και αυτή μόνο χάρη σε μια επιστημονική μέθοδο, σε μια μέθοδο στηριγμένη σε πραγματικές διαπιστώσεις μπορεί να εξασφαλιστεί. Για να είμαστε σαφείς λοιπόν. Και θα πρέπει βέβαια η προσέγγιση που θα υιοθετήσουμε να είναι και εφαρμόσιμη. Απλά εφαρμόσιμη, χωρί δυσκολίε. Θα πρέπει να λειτουργεί δηλαδή σε καθημερινή βάση χωρί δυσκολίε. Και όλα αυτά βεβαίω υπό την προπόθεση τη ε, αρχή ότι υπάρχει ανταπόδοση στη δαπάνη. Δηλαδή κόστους και αποτελεσματικότητας. Δηλαδή πρέπει και η ε, ζωή του Γεωργού να είναι πιο εύκολη, να μην ταλαιπωρείται υπερβολικά, αλλά και να κερδίζει από μια νέα μέθοδο κτηνοτροφική. Όλα αυτά νομίζω ότι αποτελούν πολλά στοιχεία, πολλά ε, δεδομένα που μπαίνουν σε έναν πίνακα. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε ένα νόμο πλαίσιο, μια νομοθεσία πλαισίου, η οποία θα τα καλύπτει όλα αυτά και που θα αποτελεί και αντίγραφο της ε, κοινή νομοθεσίας για τα τρόφιμα με την έννοια ότι χαρακτηρίζει κάθε κομμάτι νομοθεσία σχετικό με την ε, ασφάλεια των τροφίμων η νομοθεσία για τα τρόφιμα, θα πρέπει να έχουμε και το αντίστοιχο στο θέμα της κτηνοτροφίας. Αυτό πιστεύω θα πρέπει όμως να το δούμε και στις σχέσεις μας με τις τρίτες ε, χώρες. Στην Ευρώπη δεν αμφισβητεί κανείς τις προδιαγραφές ασφαλείας στα τρόφιμα διότι ε, ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές για κάθε τροφή που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ίδιο λόγο, για την ίδια αποτελεσματικότητα και διαφάνεια πρέπει να ισχύει και σε κάθε τροφή που εισάγεται από τις τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να ισχύει λοιπόν και στο θέμα της ευημερία και προστασίας των ζώων. Τώρα επισημαίνω για να επανέλθω στο κείμενό μου ότι έχω μόνο τέσσερις σελίδες περιθώριο και άρα προφανώς ε, πολλά ε, κόλπα χρειάστηκε να μετέρχομαι ή να μετέλθω για να μπορέσω να ε, καλύψω θέματα που με ενδιαφέρουν χωρίς να χάσω από την έκταση του κειμένου. Στο σημείο 5 παραδείγματι μπορεί να διαβάσει κανείς ε, πίσω από, τις, ε, πίσω από τα γράμματα την έννοια της απαγόρευσης των αντιβιωτικών στα ζώα. Επίση, στο θέμα τη σήμανση, ε, υπάρχουν διάφοροι τύποι σήμανση, διάφορε μέθοδοι σήμανση και καλό θα ήταν να ασχοληθούμε πάνω απ' όλα με τις νέες τεχνολογίες και να δούμε αν υπάρχουν δυνατότητες, φερειπίν μέσω εφαρμογών σε εφή τηλέφωνα, smartphones, ε, να λύσουμε το θέμα της σήμανσης ή της επισήμανσης ή εάν μπορούμε το ηλεκτρονικό εμπόριο να το προωθήσουμε χωρίς παράλληλα να ε, περιστέλλεται το δικαίωμα για πληροφόρηση για ενημέρωση του καταναλωτή. Από την άλλη θα πρέπει να είναι και κάτι το απλό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι πάνω σε ένα ε, πακέτο, μια συσκευασία που θα κληθεί να διαβάσει ο αγοραστής, ο καταναλωτής, δηλαδή θα υπάρχουν μυριάδες ε, διαφορών συμβόλων που δεν θα είναι ευανάγνωστα. Επίσης θα σας καλέσω να σκεφτείτε λίγο τι σημαίνει η ε, όποια πρόταση για την καθημερινή ζωή του Γεωργού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε στον δυνατόν πιο σαφείς και απλοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ να είστε όσο γίνεται πιο λίγο μίλητοι, γιατί πρέπει να τελειώσουμε στις 6.30. Η ε, Λίζαμπετ Γέγκλε και μετά ο Εβάνης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την κυρία Πάουλσεν, την συγγετρία, η οποία είπε στο τέλος την πιο σημαντική φράση που περιγράφει αυτό που κάνουμε εδώ. Ότι δηλαδή πρέπει να αναλογιζόμαστε πάντοτε τι συνέπειε έχουν οι αποφάσει μα σε αυτού που καλούνται να εφαρμόσουν την νομοθεσία, δηλαδή του γεωργού. Χωρί του γεωργού δεν μπορούμε να έχουμε καμιά επιτυχία, άρα χρειάζεται η δική του σύμπραξη. Η προσέγγιση σα μου φαίνεται καλή. Ξέρω ότι έχετε καταβάλει μεγάλε προσπάθειε για να διατυπώσετε αυτέ τι προτάσει. Και Επίσης, ε, βεβαίως προσπαθούμε να περιλάβουμε τα πάντα μέσα σε μια έκθεση, αλλά αν δεν τα καταφέρνουμε μπορούμε να συμπληρώσουμε με τροπολογίες, φαντάζομαι. Πολύ σημαντικό. Είναι η απέτηση για την προστασία της εφημερίας των την προστασία και την εφημερία των ζώων, να στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα μένα και ταυτόχρονα να υπάρχει επαρκής ασφάλεια δικαίου. Αυτό καταγράφεται στην έκθεση και είμαι ικανοποιημένη. Πολλές φορές επίσης αναφέρεται ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται έλεγχος στην υλοποίηση του δικαίου. Και εδώ βέβαια Και εδώ βέβαια η υλοποίηση, η, η εκτέλεση των αποφάσεων έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Άλλωστε βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία είχε το θέμα αυτό ως προς τους, ε, την εκτροφή πουλερικών παραγωγών ε, ορνήθων ε, μέσα από κλουβούς. Μια άλλη γραμμή πολύ σαφής που, γραμμή πολύ σαφής που διαπιστώνω στην έκθεση σας είναι αυτή που έχει να κάνει με το θέμα που συζητούσαμε και νωρίτερα, δηλαδή τις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εισαγωγή προϊόντων. Συμφωνώ απόλυτος με την προσέγγισή σας. Και επίσης ε, στις γραπτές δηλώσεις στις, ε, στα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας απευθύνουν οι ε, αγωνιστές για τα δικαιώματα των ζώων, βλέπουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος, και γι' αυτό απευθύνω έκκληση προς τους συναδέρφους, να επηρεαστούμε ιδιαίτερα από τη μία πλευρά μόνο. Γι' αυτό παρακαλώ, παρακαλώ με ψυχραιμία να εξετάσουμε τα τεχνολογικά, τα επιστημονικά δεδομένα και πάνω σε αυτά να στηρίξουμε τις προτάσεις μας και το κείμενο στο οποίο θα καταλήξουμε τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Και τελικά θα δώσω και τροπολογίες. Ευχαριστώ, Evans και μετά Ρόλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Πόλσεν και για τη δουλειά που έχει κάνει, αλλά και για την προθυμία με την οποία κάνει τις προσπάθειές της προκειμένου να καταλήξουμε σε καινή θέση για αυτό το θέμα. Είναι πολύ επικοδομητική η στάση της και ο τρόπος που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα μαζί της. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα με την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζών και ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή της στην πράξη. Η κυρία Πόλσον μίλησε για την ανάγκη να σκεφτούμε τους ε, γεωργούς. Πράγματι, υπάρχουν προβλήματα κάθε φορά που δεν εφαρμόζεται σωστά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το ξέρω κι εγώ και με τις ε, ε, όρνηθες κλοβών και με άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτό το θέμα λοιπόν της ε, θέσης εφαρμογή της νομοθεσίας είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε μια οριζόντια νομοθεσία και η ομάδα μου το στηρίζει αυτό. Η προτεραιότητά μας λοιπόν είναι καλύτερο σύστημα θέσης εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το ξέρει έγκαιρα κατά πόσο τηρούν τις προθεσμίες στα κράτη-μέλη και να φροντίζουν να αναλαμβάνουν δράση. Αυτό σημαίνει έλεγχο και καλή αντιμετώπιση έτσι ώστε οι χώρες που παραβιάζουν την νομοθεσία ή δεν την εφαρμόζουν καλά να μπαίνουν πάλι στο σωστό δρόμο. Έρχομαι τώρα στο θέμα της μεταφοράς των ζώων. Γνωρίζω ότι η σχετική έκθεση θα συζητηθεί και αυτή. Θέλουμε όμως να υπάρχει μνήα και στη μεταφορά των ζώων όσον αφορά την ε, ε καλή μεταχείριση των ζώων. Θέλουμε να υπάρχει καλή μεταχείριση των ζώων και σε προγράμματα ε, δευτέρου πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής και στη στρατηγική 2020 ενώ μέχρι τώρα μόνο 9 ε, χώρες από τις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρησιμοποιούν το θέμα, το κριτήριο της καλής μεταχείρισης των ζών στον πυλώνα 2 για πληρωμές. Τέλος, για να μιλήσω για τους γεωργούς στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια, αυτό που ακούω από αυτούς πολύ συχνά είναι ότι θέλουν ίδιες ψηλές ε, προδιαγραφές να ισχύουν και για τα ζώα τα οποία εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ζητάμε δηλαδή από τους δικούς μας τους γεωργούς να τηρούν αυτές τις προδιαγραφές, πρέπει να τις απαιτούμε και από τους άλλους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε δίκαιες και σωστές προδιαγραφές, αλλά οι γεωργοί θεωρούν ότι είναι αδικία να έρχονται προϊόντα ζώα δηλαδή απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανταγωνίζονται τα δικά τους ενώ έχουν εκτραφεί με άλλες προδιαγραφές χαμηλότερες. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους ε, κτηνοτρόφους οι οποίοι τηρούν τις υψηλές προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Εύανς. Ούρικ και μετά ο Λάιον. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εξ ονόματος του Τάνσια Ζαβού, στον ιστή της ομάδας μου, που δεν μπορούσα να είναι σήμερα παρόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πάουλσεν για το ε, σχέδιο στο θερμά και ιδιαίτερα για την ε, καλή διάθεση που έδειξε. Γιατί ε, κάλεσε εγκαίρως και προώρα, πρόημα τους ε, σκιώδεις συζητητές να συμμετάσχουν στη διαδικασία απόψεις απόψεως κτλ. Συμφωνούμε λοιπόν με την έκθεση. Αποτελεί μια καλή βάση εκκίνησης ε, για να διατυπώσουμε μια σαφή θέση για τη στρατηγική για την προστασία των ζώων 2012-2015. Και ως εκ τούτου πρέπει να μεριμνήσουμε η στρατηγική για την προστασία των ζώων να καλύπτει όλα τα ζώα και όχι μόνο τα ζώα κτηματροφικής παραγωγής. Θα πρέπει να καλύπτει και τα ζώα ε, τα οικόσιτα. Επίσης στα αδέσποτα που θα πρέπει επίσης να καλύπτει ε, το θέμα της ε, στήρωσης των ζώων αυτών πρέπει να αποτελέσει κομμάτι της στρατηγικής. και καθώς δεν καλύπτονται μέχρι τώρα από την υφιστάμενη στρατηγική θα πρέπει να τα καλύψουμε και αυτά. Τα δαϊκόσιτα, τα ζώα ζωολογικού κήπου, άλλα ζώα που μπορούν να καλυφθούν από ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με ε, ανταλλαγή πληροφοριών, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση για την προστασία των ζώων μπορούν βάσει της εκθέσεως του 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, αντιμετωπιστούν μέσα σε πολύ καλές ε, συνθήκες. Πρόκειται για ένα δίκτυο το οποίο καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο ορισμένα, όπως ακούστηκε νωρίτερα από την Επιτροπή. Η κυρία Ζάμπου λοιπόν υποστηρίζει τις προτάσεις για την προστασία των ζώων και υπογραμμίζει ότι αυτή πρέπει να καλύπτει κάθε ζώο κτηροτροφίας, αδέσποτο, οικόσιτο ζώο ζωολογικού κήπου. σαντισμής βαρός των ζώων δεν επιτρέπονται, ούτε έχουν θέσει γεωργικές εκμεταλλεύσει, οι οποίες βεβαίως εάν θέλουν να, εάν πρόκειται να είμαστε ε, αποτελεσματικοί στην ε, πολιτική μας θα πρέπει και αυτές να τηρούν τις βασικές αρχές της ευημερίας των ζώων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Λάιον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο Πόλσον για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Κάτι που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι είναι ότι πραγματικά πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στο πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει επιβολή και συμμόρφωση με την νομοθεσία που φτιάχνουμε εδώ από όσο βλέπουμε για την οδηγία για τα αυγά, τις, τις κλωβούς, είναι ότι τα κάτι μελη είναι σχετικά χαλαρά για την ομοθεσία που περνά εδώ. Και παρότι δίνουμε 10 χρόνια περιθώριο για να συμμορφωθούν, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και αν δεν συμμορφωθούν, μέχρι η Κομισιόν να προβεί στις απαραίτητε ενέργειε, να συλλέξει τις αποδείξει και να πάει στα δικαστήρια, μπορεί να περάσουν και ακόμα 3-4 χρόνια. Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή η Κομισιόν να ενεργήσει γρήγορα θα επιτευχθεί η νομοθεσία, πράγμα το οποίο καθιστά τις σχετικές νομοθεσίες αστείε. Γιατί εντάξει, περνάει η νομοθεσία, λέμε ναι, αυτό πρέπει να γίνει και μετά κανεί δεν νοιάζεται. Αυτό είναι ο τομέα που θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή. Είναι αλήθεια και για την ε, νομοθεσία περί μεταφορά των ζώων. Δεν έχει νόημα να βγάζουμε νέου νόμου από τη στιγμή που δεν εφαρμόζονται. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε και η ιδέα των ε, ορίων, ας πούμε, των ε, σημείων όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναφέρουν το τι έχει γίνει, το τι έχουν επιτύχει, όπως γίνεται με την οδηγία για τις ΟΤΟ και σώνεθες, ήταν πολύ δύσκολο το να πούνε τι συνέβη. Αν λοιπόν μπει μια απέτηση εδώ, ώστε να γίνονται αναφορές, να γίνονται έγκαιροι έλεγχοι, επιθεωρήσεις, μπορεί να υπάρξει κάποια πρόοδος. Επίσης να προβλέψουμε κυρώσεις μέχρι την τελική ημερομηνία εφαρμογής της νομοθεσίας. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες και ποια θα είναι η νομική βάση ώστε η Κομισιόν να μπορεί όντω να προβεί σε εγκαιρή δράση και αντί να προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν ενώ έχει περάσει η προθεσμία και πολύ μετά, καλύτερα είναι να βρούμε τρόπους ώστε όλοι να συμμορφώνονται στην κατάλληλη προθεσμία. Νομίζω πως αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στις προτάσεις. Κατά τα άλλα συμφωνώ με την κατεύθυνση που έχετε ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Η Μπρίτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την πολύ εντατική συζήτηση που μπορέσαμε να αναπτύξουμε και πριν από δύο τύπους του εγγράφου και όχι μόνο οι αλλά και όλοι όσοι ενδιαφέρθηκαν για το κείμενο. Θα ήθελα να αναφερθώ στο δικαίωμα για ενημέρωση του καταναλωτή. Ε, θα υπογραμμίσω εδώ ότι έχει σημασία όχι μόνο για τον γεωργό, αλλά και για τον καταναλωτή. Το δικαίωμα στην ενημέρωση είναι σημαντικό όχι μόνο ως μονόδρομος, δηλαδή να λέει ο καταναλωτής έχω δικαίωμα στην ενημέρωση, αλλά να επιδιώκει να λάβει την πληροφορία, να μην είναι δηλαδή μονόδρομος, αλλά ε, αμοιβαία σχέση αυτή. Συμφωνώ κατά τα άλλα ότι θα πρέπει η προσία των ζώων να στηρίζεται και όποιο μέτρο εισαχθεί θα πρέπει να στηρίζεται σε ε, επιστημονικά μέτρα και ότι θα πρέπει να επηρεαζόμαστε από τα μερικές φορές ε, ιδιαίτερα συγκινητικά γράμματα που λαμβάνουμε, email κτλ. Συγκινητικά μέχρι και ε, απειλητικά μερικές φορές. Εν πάση περιπτώσει όμως πρέπει ψύχρεμα να λάβουμε μια απόφαση. λαμβάνοντας υπόψη και τι θα σήμαινε το να μην βρεθεί λύση, γιατί ε, το να μην υπάρχει επαρκής ρύθμιση θα σήμαινε ταυτόχρονα και στρέβλωση ανταγωνισμού. Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχει κάποια δυνατότητα στα κράτη-μέλη στα οποία διαπιστώνεται ότι υπάρχει ε, στρέβλωση ανταγωνισμού λόγω της μη εφαρμογής ε, ε, της νομοθεσίας, μη σωστής εφαρμογής νομοθεσίας, να απαιτείται και κάποια επιστροφή ε, οικονομική ε, για να υπάρχει αυτή η αντιστάθμιση σε με αυτούς που έχουν χάσει, έχουν υποστεί κάποια οικονομική επιβάρυνση λόγω της αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας. Και άρα ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάποια ποινή, ούτως ή διότι υπάρχουν κράτη τα οποία, όπως είπα, για να εξασφαλίσουν ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς τους δεν εφαρμόσουν σωστά την ε, νομοθεσία, ενώ υπάρχουν άλλα τα οποία είναι πιο αυστηρά ακόμη από την εφιστάμενη νομοθεσία. Ε, δεν θα έπρεπε ίσως να δεχθούμε να υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι συνθήκες διαβίωσης, προστασίας, μεταχείρισης δεν μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ε, πόσα ζώα έχει κανείς ε, στην ε, εκμετάλλευσή του. Θα πρέπει πάντοτε να είναι οι συνθήκε τέτοιε, βέβαια προσαρμοσμένε στι συνθήκε εκτροφή, ανάλογα με την εκμετάλλευση, ώστε το ζώο να μην υποφέρει. Θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε πιστοποιητικά. Ε, εάν διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη να προσφέρετε κατάρτιση στον κτηνοτρόφο. Αν και πρέπει να πούμε ότι μερικοί από τους γεωργούς μας έχουν πάρα πολύ υψηλή κατάρτιση, ε, ε, μέχρι και μεταπτυχιακό ορισμένοι από αυτούς και ίσως εκεί αποδεικνύεται περιττό το επιπλέον πιστοποιητικό. Άρα, ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κατάλογο που θα πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς σπουδών στην Ευρώπη που ε, θεωρείται ότι είναι επαρκής και ότι καλύπτουν αυτήν την ανάγκη για το πιστοποιητικό. Ιδιαίτερα για αυτούς τους γεωργούς που έχουν επαρκή κατάρτιση όπως έλεγα. Και επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε τις υπερβολικές ρυθμίσεις. Διαπιστώνεται άλλωστε ότι πολύ συχνά είναι και αντιφατικές μεταξύ τους οι ρυθμίσεις, φερειπίν στη μεταφορά ζών των ζώων Ε, και θα θυμηθώ το παράδειγμα ενός ε, παραγωγού ηχθειοτρόφου, ο οποίος μου είχε διαμαρτυρηθεί γιατί έλεγε ότι η νομοθεσία περί μεταφορά ζώων τον υποχρέωνε όταν ήθελε να μεταφέρει τις πέστροφές του ε, μέσα σε δεξαμενές με νερό κτλ. να τις ποτίζει πότε πότε. Οπότε φαντάζεστε ότι το φαινόταν λίγο δύσκολο αυτό το πότισμα της πέστροφας. Εν πάση περιπτώσει α μην κάνουμε και υπερβολικές ρυθμίσεις, παραμένουμε λογικοί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέρλινγκ. Και συγχαρητήρια, κατέστητε τακτικό μέλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα για αυτή την έκθεση και να τονίσω ότι δεν είμαι επίσημο και όδηση ηγητή εδώ, αλλά θα τα πω αυτά με την ιδιότητα της Ευρωβουλευτού. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως πρόκειται για μια στρατηγική και συγχαίρω την εισηγήτρια γιατί είναι πάντα πολύ δύσκολο να μείνει κανείς στα στρατηγικά ζητήματα και να μην χαθεί στις λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχουν ένα-δύο τομεί όπου πιστεύω θα έπρεπε να είμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι. Το πρώτο είναι αυτή η ε, αυτός ο τονισμός της επιβολής. Το, το είπαν όλοι και το επαναλαμβάνω και εγώ. Ίσως θα πρέπει να πούμε πρώτα ποιες είναι οι οδηγίες οι οποίες ε, δεν έχουν ε, ακόμα εφαρμοστεί πλήρως. Δεν χρειάζεται να τις αλλάξουμε αυτές, απλώς πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Και θα ήθελα αυτό να αναφερθεί, ας πούμε αυτή για τους ολογικούς σκήπους, παράδειγμα. Επίσης πρέπει να λάβουμε απόφαση για το κατά πόσο θέλουμε να συμπεριλάβουμε εδώ τα δέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ίσως θα είναι θέμα ε, κρατών μελών και όχι θέμα ευρωπαϊκό. Υπάρχουν βέβαια προτάσεις για να να, να αφαιρεθούν από εδώ αυτά τα ζώα, αλλά το, η αναφορά στο kept animals ε, ε, ζώα υποκράτηση δηλαδή, υπό περιορισμό θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Τώρα, Επίσης θα πρέπει να θυμηθούμε τη δέσμευση του Επιτρόπου Ντάλι κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας ε, και τη σχετική συζήτηση εκεί για την ενημέρωση για τα τρόφιμα για τους καταναλωτές. Οπότε αυτό το θέμα του είδους της φαγής στην ουσία αφέθη κατά μέρος επί τη βάση του ότι θα μιλούσαμε γι' αυτό, θα μιλούσε γι' αυτό ο Επίτροπος μέσα στη στρατηγική για την ε, ευημερία των ζώων. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε τι ακριβώς κάνει η Κομισιόν για αυτό το θέμα και πού ακριβώς θα ενταχθεί το ζήτημα αυτό, γιατί δεν έχουν δοθεί και πολλές λεπτομέρειες για όλο αυτό. Και ήταν μια συγκεκριμένη δήλωση από το σύνολο των επιτρόπων ότι θα καλυφθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα υποβάλω λοιπόν σχετική τροπολογία για να καλυφθεί το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Τζούλη, ευχαριστούμε και τώρα δίνουμε το λόγο στην Κομισιόν. Α, ο Μισελ έχει ζητήσει το λόγο, συγγνώμη. Δεν σας είδα. Ναι, Πρόκειται για ένα θέμα που δεν είναι το ίδιο ε, ευαίσθητο σε όλες τις χώρες. Ωστόσο πρόκειται για μια στρατηγική, για ένα πρόγραμμα πλαίσιο δηλαδή και σημειώνονται στην έκθεση γίνεται η σχέση, ο συσχετισμός ανάμεσα στην ευημερία των ζώων και την δημόσια υγεία. Υπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες για να εξετάσει κανείς την ευημερία των ζώων. Εγώ θα ήθελα να προσθέσουμε ένα σημείο στην στρατηγική που θέλει να φτιάξει η Κομισιόν το θέμα της κατάστασης υγείας των αγρίων ζώων. Που ένα και ποιος να ε, συγχροντίζεται με τα κατοικίδια ζώα. Σε κάποια κράτη επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι ανάμεσα στα άγρια ζώα αναπτύσσονται αρρώστιες, ασθένειες οι οποίες είναι μεταδοτικές και μπορεί να μεταδοθούν στα κατοικίδια ζώα αλλά και στον άνθρωπο. Και η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ενδιαφέρεται και για αυτό το ζήτημα γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ευημερία των ζώων. Σα ευχαριστώ, Μισελ. Το λόγο έχει τώρα η Κομισιόν, ο δόκτωρ Σιμονίν. Παρακαλώ και μετά κλείνουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Ε, η συζήτηση είναι ευρύτατη. Απλώς θα ήθελα να κάνω κάποιες ευκρινήσεις για κάποια σημεία που νομίζω ότι θα μπορούσαν να αποσαφηνιστούν καλύτερα όσον αφορά τους σκύλους και τις γάτες ή τα ζώα συντροφιάς, αλλά πιο συγκεκριμένα σκύλοι γάτες. Είναι ενδιαφέρον ε, ότι έγινε σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο στα τέλη του 2010 υπό την Βελγική Προεδρία και ζητήθηκε από την Κομισιόν να προβεί σε διάφορες μελέτες για τα ζώα, τους σκύλους και τις γάτες ε, που είναι αντικείμενο εμπορίας. Ε, μέσα σε αυτή τη στατικική προβλέπεται μελέτη ακριβώς για την σκοπιμότητα ή όχι της λήψης μέτρων στον τομέα αυτό να επιστήσω ωστόσο την προσοχή των Ευρωβουλευτών ότι όσον αφορά τα εγκαταλελειμμένα ζώα, δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε αρμοδιότητα εμεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα ευημερία σε αυτόν τον τομέα σε κάποιε χώρε, αλλά είναι επίση αλήθεια πω υπάρχει και πρόβλημα αρμοδιότητα με βάση τη συνθήκη, γιατί είναι σημαντικό αυτό να το υπογραμμίσουμε. Το άρθρο 13 της συνθήκης δεν δίνει εντολή στην Ένωση για να ασχοληθεί με θέματα ευημερίας, αλλά απλά ζητά να τα λάβουν υπόψη πόσον υπάρχουν ε, στόχοι της Ένωσης οι οποίοι τίθενται σε εφαρμογή. Ε, κάτι ακόμα που θέλω να υπογραμμίσω γιατί είναι κάτι το οποίο συγκεκριμένα αναφέρθηκε είναι η δικαιοθεσία όσον αφορά την ε, ζάλη των ζώων είναι, έχει αναλάβει η Κομισιόν ε, την ε, υποχρέωση να, κάνει μια μελέτη ε, για τον τρόπο θανάτωσης των ζώων και την σχετική ετικετοθεσία. Αυτό είναι μέσα στο κατάλογο δράσεων που έχουν προσαρτηθεί στη στρατηγική. Σας ευχαριστώ. Το τελευταία λέξη έχει αντιπρόεδρος Φόλσον. Πρόεδρε, βεβαίω όλα τα ζώα θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα νομοπλαίσιο. Εδώ όμως αναφέρομαι ιδιαίτερα στα ζώα της κτηνοτροφίας για τον λόγο ότι αυτά είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των ζώων Και για τα αδέσποτα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τα φτάσουμε δεδομένου ότι είναι αδέσποτα ακριβώς, δεν είναι κάπου σε έναν ελεγχόμενο χώρο, έτσι δεν είναι. Να σας πω, και εγώ μένω σε μια περιοχή κοντά σε δάσους και είδα τι ε, προάλλες ε, μια γεριλίκο να έχει αρπάξει μια άλκη. 300 μέτρα από το σπίτι μου, από το παράθυρό μου το είδα. Ε, τι θα κάνω νομοθεσία και γι' αυτό. Μην ξεχνάμε, η νομοθεσία για τι οτόκε όρνηθε είχε περάσει μέσα από μια διαδικασία 12 ετών προετοιμασία και η Επιτροπή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να αλλάξουν ένα κόμμα πριν περάσουν τα 12 χρόνια, ακόμα και σε περίπτωση παράβασης καρών από τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός νομικός, ο οποίος θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρεί τον έλεγχο μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Για δε την επισήμανση, θα ήθελα να πω ότι ναι, είναι χρήσιμη η επισήμανση, αλλά εφόσον είναι ορθή εφόσον ευσταθεί. Διότι υπάρχει νομοθεσία για την σφαγή των ζώων, την προετοιμασία του για τη σφαγή κτλ. με συγκεκριμένε εξαιρέσει. Δεν θα ήταν όμως πιο σημαντικό να εφαρμοστεί η φυστάμενη νομοθεσία πάνω απ' όλα και να μεριμνούμε στο να γίνεται η των ζώων πριν από τη σφαγή. Γιατί είναι πολλέ οι χώρε που μεγάλο ποσοστό, συντριπτικό ποσοστό των ζώων, 80% των ζώων δεν αναισθητοποιούνται πριν σφαγούν. Παρότι υπάρχουν οι κανόνε. Παρότι θα ήταν υποχρεωμένο να το κάνουν. Άρα, σα ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ήταν πραγματικά καταπληκτική συζήτηση. Πολύ καλή δουλειά κάναμε μαζί με του συντονιστέ και όλου του συναδέλφου που εξέφρασαν το ενδιαφέρον. Σα ευχαριστώ θερμά όλου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και υπενθυμίζω ότι έχουμε προθεσμία τις 30 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι για την κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ τους πάντες. Έληξε το συνεδρίαση της Επιτροπής μας και αύριο το πρωί ξεκινάμε με τους συντονιστές στις 9, στις 10 παρατέταρτο με την Ολομέλεια της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ θερμά και καλή σας βραδιά.